Uh, Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε. Υπάρχει περίπου απαρτία, οπότε μπορούμε να αρχίσουμε έτσι κι ε, όσο περνάει η ώρα όλο και περισσότεροι θα μπαίνουν στην αίθουσα. Εγκρίνεται την ημερήσια διάταξη πρώτα απ' όλα. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται. Σημείο 2. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Σας ενημερώνω ότι η συνεδρίασή μας περνάει στο διαδίκτυο. Γι' αυτό για να σας ε, παίρνει η κάμερα και να φαινόσαστε στην οθόνη θα πρέπει να πατάτε το κουμπί του μικροφόνου που βρίσκεται αριστερά σας. Έχετε λάβει διάφορα σημειώματα. Ό,τι παρατηρήσεις έχετε παρακαλώ στη γραμματεία έχουμε 4 Σεπτεμβρίου συνάντηση με τον πρέσβη. Επειδή έχουμε την ετήσια διάσκεψη των επικεφαλής ε, ε, των αντιπροσωπιών εν ώψη της 7ης Σεπτεμβρίου που θα γίνει συνάντηση εδώ στις Βρυξέλλες. Οπότε την 3η 4 Σεπτεμβρίου έχουμε συνάντηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το απόγευμα θα έχει ως εξής συνάντηση. 3 με 3 και 45 ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο Σούλτς. 15.65 μέχρι τις 6 με ανταλλαγή απόψεων με τους πρόεδρους των αντιπροσωπιών. Οι εισαγωγικές παρατηρήσεις του Έλμαν Μπροκ, του Μάικλ Κάσμαν και των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Υπάρχουν και προσκλήσεις από άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ και του πρόεδρου του. Στι 6 υπάρχει μια μικρή δεξίωση από τον πρόεδρο Σούλτ. Οπότε διμερώς εκεί θα μπορέσουμε να έχουμε και άλλε επαφέ. Και εφόσον έρχεται η υπηρεσία εξωτερική δράση με 140 πρέσβει επικεφαλή αντιπροσωπιών και συμμετέχοντε, ε, επίση και από τι επιτροπέ κοινοβουλευτικέ κλπ., Μόνο οι πρόεδροι και οι αντιπρόσωποι του προβλέπονται εκεί. Γιατί 140, σε ποια αίθουσα δηλαδή θα συνεδριάσουμε, το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε ακόμα. Θα πρέπει να βρούμε μια μεγάλη αίθουσα πάντω για να χωρέσουμε όλοι. Ωραία. Κατάσταση πρόοδου των υποεξέλιξη τριμερών διαπραγματεύσεων. Σε σχέση με τον κανονισμό πλαίσιο για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ε, καταθέσει τις ε, προτάσεις τους για μακροοικονομική αρρωγή προς τρίτες χώρες. Έγινε τριμερής διάλογος στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Καζάκ είναι συγκητή για αυτό το θέμα, αλλά δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή ο Μετίν Καζάκ. Οπότε δεν έχουμε σχόλιο. Όταν έρθει θα του δώσουμε το λόγο να μας πει λίγα πράγματα. Όσον αφορά τώρα τις εμπορικέ προτιμήσεις για το Πακιστάν, εδώ πέρα υπάρχει μια πρόταση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έκτακτες διατάξεις όσον αφορά αυτό. Ο Μαρέκη ε, η συγγετή μας ε, έγινε ήδη στο Στρασβούργο μια πρώτη συνάντηση, η Δανέζικη Προεδρία ήταν παρούσα, δέχονται κάποιες από τις τροπολογίες που εγκρίναμε εμείς τον Μάιο του 2010 και αυτό που ήταν επίμαχο ήταν το θέμα των ελέγχων που αντικαθίσταται τώρα από μια πιο πλοπημένη διαδικασία προκειμένου να βγουν κάποια προϊόντα από τον κατάλογο προτιμησιακής μεταχείρισης. Το Κοινοβούλιο πάντως δεν αντιλαμβάνεται τη στάση του Συμβουλίου γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν δασμοί ή περιορισμοί στις πρώτες ε, ύλες από το Πακιστάν που χρησιμεύουν για την κατασκευή προϊόντων που καλύπτονται από τον κανονισμό. Εγώ σας τα λέω τώρα, δεν ξέρω. Εσείς τα καταλαβαίνετε φαντάζομαι καλύτερα από μένα, λέει ο Πρόεδρος. Δεν υπήρξε συμφωνία. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε μέλλον με τον τριμερή διάλογο. Σχόλια. Όχι, ε. Ευτυχώς λέει ο Σημείο 4. Τροποποίηση του κανονισμού για τη θέσπιση ενό κοινοτικού συστήματο ελέγχου των εξαγωγών τη μεταφορά, τη μεσητεία και τη διαμετακόμιση ειδών διπλής χρήση. Εδώ έχουμε τον εισηγητή. Κρίστοφερ, έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ όλους Στα σουηδικά θα μιλήσω, οπότε ετοιμαστείτε. Λέει ο μιλητή. Βάλτε τα ακουστικά σας. Λοιπόν. Μάλιστα, ποια είναι η προϊστορία το σκηνικό αυτής της πρότασης που περιγράφει την τελευταία φορά. Πρόκειται η διαδικασία για αυτούς τους καταλόγους για αγαθά με διτή, διπλή χρήση να επιταχυνθεί και να απλουστευτεί, διότι όπως επανειλημμένα έχουμε πει, σε όλη αυτή την επικαιροποίηση υπάρχουν συχνά πολλά προβλήματα σύμφωνα με την τακτική, τακτή νομοθεσία όπως προβλέπετε το νομοθετικό πλαίσιο. Για αυτή τη διαδικασία εδώ πρόκειται για χώρες ή για άτομα να υπάρχουν κυρώσεις όταν δεν έχουν συμπεριφερθεί σωστά, ώστε να μην έχουν πλέον πρόσβαση σε αυτά τα αγαθά. Δεδομένων όμως των ταχαίων εξελίξεων από τεχνολογικής πλευράς χρειαζόμαστε μια απλή διαργασία, μια ε, ταχύτερη διαδικασία ώστε να μπορούμε να επικαιροποιούμε αυτούς τους καταλόγους. Αλλά υπάρχει και μια πτυχή για τον ανταγωνισμό σε όλα αυτά, διότι υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις για αυτά τα διτής χρήση αγαθά που εργάζονται ακριβώ σε αυτόν τον τομέα. Κρίμα θα ήταν αυτοί να υποστούν τι κυρώσει επειδή κάποιε χώρε ε, είναι ταχύτερε στην επικαιροποίηση δικών του καταλόγων και διεργασιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι σημαντικό αυτή η νέα νομοθετική πρόταση το δυνατόν ταχύτερα να εγκριθεί διότι δεν υπάρχουν πολιτικέ αντιπαραθέσει ή τριβέ σε αυτό το ζήτημα. Αυτό καταδείχθηκε και από τι συζητήσει. Δεν υπάρχουν προβλήματα και σε συζητήσεις με το Συμβούλιο. Καταδείχτηκε με όλα αυτά συνολικά ότι Πρόκειται για τεχνικής, ε, τεχνικού χαρακτήρα λεπτομέρειες. Λάθος θα ήταν λοιπόν αν στο νομοθετικό έργο εμείς καθυστερούσαμε λόγω τέτοιου είδους ε, ε, τεχνικών λεπτομεριών. Κυρίως πρόκειται, και όπως αναφέρθηκε, για το ότι δεν θα πρέπει οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να υποστούν πλήγματα όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Να μην πληγεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα λόγω βραδύτερης επικαιροποίηση και εξυγχρονισμού. Το θεωρώ σημαντικό σε αυτό το έργο, αλλά επίσης και για το μέλλον να προσέξουμε σε μελλοντικές τέτοιες επανεξετάσεις και αναθεωρήσεις να μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό και πιο διαφανές πλαίσιο εργασίας. Τουλάχιστον αυτό είναι ο στόχος της εργασίας μου με αυτές τις προτάσεις. Δικό μας, δική μας δουλειά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι τους γενικούς ελέγχους, ε, να μπορέσουμε να τους διασφαλίσουμε στο αναγκαίο πλαίσιο. Όχι όμως την μικροεποπτεία για κάθε είδους ίσονο σημασία ε, τεχνικού χαρακτήρα λεπτομέρειες. Γι' αυτό όπως και την τελευταία φορά ανέφερα, η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρώ ότι είναι θετική. Το ίδιο πιστεύει και το Συμβούλιο. Αν δεν υπάρχουν κάποιες ενστάσεις από κάποιους λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε ταχύτερα και πραγματικά αυτό το, αυτή τη μικροδιαχείριση να την ολοκληρώσουμε, να την κλείσουμε από πλευρά Κοινοβουλίου και να επικεντρωθούμε στους γενικούς ελέγχους. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε, Κρίστοφερ. Φραντσέσκα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την έκθεση. Υπάρχουν δύο κύριες πτυχές εδώ. Αφενός, αναφέρεται το πρόβλημα που μπορεί να έχει ο κλάδος. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει και η πτυχή ασφάλεια του όλου ζητήματος, που νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε πολύ. Θα ήταν εφικτό να έχουμε τον κατάλογο των χωρών, έτσι ώστε να μπορεί πολύ γρήγορα να αντιδράσει σε εξελίξεις στις χώρες αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον προκύψει κάτι. Το θέμα αυτό έχει να κάνει περισσότερο με νέα όμως προϊόντα που μπαίνουν στην αγορά. Γι' αυτό εδώ πιστεύουμε ότι πρέπει να συζητηθεί ε, το θέμα και να υπάρχει δυνατότητα εξάντε να γίνονται έλεγχοι. Άρα χρειαζόμαστε τον ε, βασικό κανονισμό που να λέει ότι μπορούν να γίνονται έλεγχοι πριν εισαχθούν τα προϊόντα αυτά. Όλοι εξαρτώνται από αυτό το βασικό κανονισμό, δηλαδή κατά από ποιε προϋποθέσεις, προϊόντα ή χώρες θα μετατίθενται από τον ένα κατάλογο στον άλλον. Καλό θα ήταν να περιμένουμε λοιπόν αυτό το βασικό κανονισμό, να δούμε τι λέει πριν δώσουμε τις κατεξουδότηση πράξεις, για να ξέρουμε κάτω από τι συνθήκες παραχωρούμε τέτοιες κατεξουσιοδότηση πράξεις και μετά να αποφασίσουμε. Αυτό είναι το σχόλιο που έχουμε εμείς ως πράσινοι. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Άλλος κανείς, υπάρχουν σχόλια, όχι. Ωραία, τότε θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γκαζότη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την ε, ξέρετε δουλειά που έχει κάνει όσον αφορά αυτή την πρόταση. και για τον τρόπο με τον οποίο προχωράει αυτή η υπόθεση. Όντως είναι πολύ σημαντικός ο κανονισμός αυτός. Πριν από πέντε μέρες πρέπει να ξεκινήσει να ισχύει ο κανονισμός έτσι ώστε και οι εξαγωγείς να μπορούν να υποφελούνται από τις αλλαγές στο καθεστώς αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έχω μερικά σχόλια όσον αφορά τις τροπολογίες. Η πρώτη τροπολογία, από ό,τι βλέπω, έχει να κάνει με την πλήρη ενημέρωση και τεκμηρίωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι το κείμενο του κανονισμού πρέπει να ακολουθεί τις γενικές διατάξεις έτσι όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί στα πλαίσια του Μνημονίου για Κατανόηση. Πρέπει να μείνουμε δηλαδή σε αυτό και γι' αυτό και προτείνουμε ε, να διατηρηθεί η στάνταρ διατύπωση για την τροπολογία αριθμός 2. Πιστεύουμε ότι είναι μια καλή ιδέα, διότι δείχνει μεγαλύτερη συνέπεια έτσι όπως προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευχαρίστω θα το υποστηρίξουμε αυτό. Τρίτη τροπολογία τώρα. Εδώ. Δεν βλέπουμε να χρειάζεται μια τέτοια τροπολογία. Και ιδιαίτερα μάλιστα επειδή οι εξουσιοδοτήσεις θα ήταν καλύτερα να μένουν για την περίοδο που προτείνει η Επιτροπή. Φυσικά καταλαβαίνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει τακτικά να ενημερώνεται και τακτικά ε, να αναθεωρεί ενδεχομένω τις εξουσιοδοτήσεις. Θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτι για τα κάθε τρία χρόνια για τον κανονισμό ή να πούμε ότι η δεύτερη έκθεση θα πρέπει να γίνει στα έξι χρόνια. Κάτι τέτοιο θα μας επέτρεπε να μην πρέπει να έχουμε παρουσίαση κανονισμού κάθε τρία χρόνια και για τις εξοδοτήσεις κάθε πέντε χρόνια. Και ένα τελευταίο σχόλιο, επιτρέψτε μου, που έχει να κάνει και με την ερώτηση που βάζουν οι πράσινοι. Οι προϋποθέσεις για το ποια ε, προϊόντα μπαίνουν ή βγαίνουν από τον κατάλογο έτσι καλώς έπρεπε όλα αυτά να συνάδουν με τα προηγούμενα καθεστώτα τα οποία καθορίζουν τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών μελών. Και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχουμε. Άρα δεν υπάρχει μεγάλη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής όσον αφορά τα προϊόντα. Συμφωνούνται βάσει των καθεστώτων στα οποία συμμετέχουν οι χώρες μέλη. Και εμείς πρέπει ό,τι κάνουμε να είναι σύμφωνο με αυτά. Αυτό προς διευκρίνηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, βλέπω ότι είσαι σκιώδης, θέλεις να σχολιάσεις κάτι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και ζητώ συγγνώμη για την ελαφρά αργοπορία μου. Πέρα από την καλή δουλειά του Σκιώδους, θα ήθελα να θέσω και κάποια ερωτήματα και σε αυτόν και ε, στην Κομισιόν. Το πρώτο μου ερώτημα αφορά τη διαδικασία. Υπήρξε ε, διαβούλευση επί πράσινης βίβλου με προθεσμία την 31η Νοεμβρίου του 2011 ε, και βλέπω ότι δεν υπάρχει καμία συνέχεια από αυτού και αυτό με ανησυχεί γιατί περνάει ο χρόνος και ξέρουμε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις ε, είναι πολύ γρήγορες και το Κοινοβούλιο ορθώς έχει καταδείξει επανειλημμένα ότι οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ γρήγορες και ε, ε, όταν οι διαδικασίες μας δεν προσαρμόζονται αντίστοιχα χάνουμε χρόνο διότι η κατάσταση εξελίσσεται λοιπόν θα ήθελα να το σχολιάσω Επίσης η επικαιροποίηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ενδεχομένως ε, και την πλήρωση κενών θέσεων που από ό,τι, από καταλαβαίνω στην Κομισιόν ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Επίσης, κατηγοριοποίηση κάποιων από τις τεχνολογίες που αναφέρονται. Ε, θα ήθελα όμως ε, να μου πούν εάν υπάρχει χώρος και για κατηγορία η οποία θα μπορούσε να είναι single use μίας χρήσης που ε, μπορούν ε, να οδηγήσουν σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ε, νέα μηχανήματα τα οποία ακριβώς χρησιμοποιούνται για δίωξη, για παρακολούθηση κτλ. Και επομένως ξέρουμε από μαρτυρίες φυλακισμένων ε, ότι ε, διεπίστωσαν ότι υπήρχε καταγραφή όλων των ηλεκτρονικών τους μηνυμάτων, των ε, επικοινωνιών που είχαν μέσω του κινητού τους τηλεφώνου κτλ. Ε, και όλα αυτά καθίστανται δυνατά μέσω εξαγωγής προϊόντων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποιο τρόπο ε, να δημιουργήσουμε κατηγορία των προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο ε, για την καταστολή ιδεών ανθρώπων κτλ. Τελική ερώτηση. Εφαρμογή και αξιολόγηση μαθαίνουμε, διαβάζουμε, το ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα πεδίο διαρκώς ε, ε, μεταβαλλόμενο. Επομένως αυτά που ισχύουν τώρα ίσως δεν ισχύουν τον επόμενο μήνα. Υπάρχει σκέψη για αξιολόγηση ε, τεχνολογικών τομέων τρίτων χωρών και επίσης τι γίνεται με την επιβολή ας πούμε των ε, κανόνων για την ώρα δεν βλέπουμε να υπάρχουν κυρώσεις. Οι κυρώσεις κατά κανόνα ε, αφορούν τις χώρες μέλη. Ε, μήπως πρέπει να προβλεφθούν ε, ε, ισόρροπες κυρώσεις για όλες τις πλευρές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σάκα. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, όταν έγινε η χαρτογράφηση ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, είδαμε ότι είχαμε πάρα πολλές περιπτώσεις σπασίματος των υπολογισμών, hacking. Είναι γεγονός ότι πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Κρίστοφερ, θέλεις να πάρεις το λόγο μια και δεν επιθυμεί κάποιος άλλος και μετά στην Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. για τη, διπλή χρήση. Για την ε, διπλή αυτή χρήση, λοιπόν. Επίσης και για το θέμα πώς θα διαμορφωθεί η συνέχεια για το πράσινο βιβλίο. Εν πάση περιπτώσει δεν θα επαναλάβω αυτά, αλλά κάποια πράγματα που συμφωνώ μαζί σας. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ένα πράγμα, διότι πολλά ενδιαφέροντα θέματα τέθηκαν για τη διπλή χρήση, τον κανονισμό για τη διπλή χρήση. Θα εξετάσουμε το σύνολο της διπλής χρήσης ως σύστημα εν ευθέτω χρόνο. Όμως σε αυτή την έκθεση επικεντρωνόμαστε σε ένα κύριο θέμα. Να μεριμνήσουμε να υπάρχει μια ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή και υλοποίηση. Διότι έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Η, το ένα θέμα μιας τεχνολογίας κάποια χρονική στιγμή μπορεί να έχει τελείω διαφορετική όψη υστερότερα. Γι' αυτό και έχουμε και το καλύτερο επιχείρημα υπέρ τη ε, προσέγγιση μα. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε την κανονική νομοθετική διαδικασία για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Επίση πρέπει να είμαστε πιο ταχής και αποτελεσματική. Υπάρχει κάποια διαφορά εδώ σε σχέση με την τεχνική, ας το πω έτσι, ε, συνιστόσα. Από την άλλη πλευρά χρειαζόμαστε ταχύτατα τον γοργό χαρακτήρα του πίνακα του καταλόγου αυτού για να είμαστε αποτελεσματικοί. Λοιπόν, πολλά σημαντικά θέματα θίγεται για το θέμα του κανονισμού διπλής χρήσης. Ελπίζω ότι υστερότερα θα μπορέσουμε μεταγενέστερα να επανέλθουμε σε αυτά. Εδώ θα ήθελα όμως να επικεντρωθούμε σε μια ταχεία διαφανή διαδικασία για τη διευθέτηση αυτών των θεμάτων. Ήθελα να το τονίσω αυτό. Δεν ξέρω, ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επανέλθει για κάποια από τα θέματα που τέθηκαν, που προφανώς στοχεύουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν είχαν καλυφθεί. Ίσως με μια δεύτερη προσπάθεια μπορούμε να τα καλύψουμε. Uh, Thank you, sir. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι βεβαίως ε, καλωσορίζουμε οποιαδήποτε βοήθεια για πλήρως κενών θέσεων στην Κομισιόν ε, και πρέπει να σας πω ότι για αυτό το θέμα ε, της ε, διπλής χρήσης. Ε, έχει υπάρξει κάποια πρόεδρο σε σχέση με την πράσινη βίβλο. Ε, κυρίως όσον αφορά την επιβολή και την αξιολόγηση. αυτό είναι το κύριο ζήτημα το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μέσω της πράσινης βίβλου. Θέλαμε δηλαδή να ε, δημιουργήσουμε μια βάση διαβουλεύσεων, βάση της οποίας η Κομισιόν ε, θα μπορεί να προωθεί σε εσά την έκθεση για την ε, υλοποίηση και το βαθμό υλοποίηση του κανονισμού, έτσι ώστε να υπάρξουν και νέες προτάσεις προς κάθε κατεύθυνση. Στην Πράσινη Βίβλο ε, προβλέπεται και ε, πιο κοινή αντιμετώπιση του θέματος της ε, υλοποίησης και της εφαρμογής της αδειοδότησης των εξαγωγών, δηλαδή την χορήγηση αδειών εξαγωγής λοιπά. Επίσης, αυτό που σαφώς αναφέρεται στην πράσινη βίβλο είναι ότι είμαστε νέα αγορά και αυτό ισχύει και για τα προϊόντα διπλής χρήσης και είναι γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιοι, να υπάρχουν μάλλον κάποιες ε, ε, διαστάσεις όσον αφορά τις ε, εξαγωγές. Απ' την άλλη πλευρά, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθούν κάποια προϊόντα από κακόβουλους ανθρώπους με κακόβουλες προθέσεις, αλλά από την άλλη πλευρά βεβαίως πρέπει να βοηθήσουμε και τους εξαγωγείς μας. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, πριν το τέλος του τρέχοντος έτους πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια τελική έκβαση του, ε, της ε, ε, συνέχειας που θέλει η Κομισιόν να δώσει στην Πράσινη Βίβλο και επομένως να έχουμε κάποιες και μετά να έχουμε μια περιοδική έκθεση κάθε τρία χρόνια. Όπως είπα, ε, υπάρχει χώρος βάσει του κανονισμού έτσι ώστε οι χώρες να ελέγχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ε, οπωσδήποτε πάντως ε, θα συζητηθούν ε, όλα τα στοιχεία και θα συνεκτιμηθούν οι απόψεις, αλλά βεβαίως τα κράτη-μέλη θα έχουν την τελική διακριτική ευχέρεια για απόφαση, ενώ η πράσινη βίβλος θα δώσει την απαραίτητη πολιτική καθοδήγηση και βεβαίως θα συλλέξει οι απόψεις όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων όσον αφορά την ε, ε, γρήγορη εξέλιξη της τεχνολογίας. Ορθώς λέει ο μιλητής ε, ότι γι' αυτό θέλουμε αυτόν τον κανονισμό έτσι ώστε να μπορούμε να τροποποιήσουμε τα παραρτήματα και δύο και τρεις φορές το χρόνο και όχι μονάχα μία φορά κάθε δύο χρόνια έτσι όπως προβλέπετε στην τωρινή εκδοχή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ προθεσμία υποβολής τροπολογιών 22 Ιουνίου 12 το μεσημέρι, 11-12 Ιουλίου η έγκριση της έκθεσης, ψήφος ή στην Ολομέλεια, στην Σύνοδο του Νοεμβρίου. Άψογα, προχωράμε λοιπόν. Αντιπροσωπεία ad στην Κολομβία και το Περού. Δυστυχώς και οι δύο υπεύθυνοι δεν είναι εδώ. Ε, απουσιάζουν, επομένως προτείνω αναβολή μέχρι της αφήξεώς τους. Σημείο 6. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ σχετικά με την συμμόρφωση και την αποδοχή των βιομηχανικών προϊόντων ΔΣΑ και πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας. Από ό,τι φαίνεται έχουμε πλέον συμφωνία. και αναρωτιέμαι ποιο θέλει να μιλήσει, να πάρει το λόγο από τις ε, πολιτικές ομάδες. Δεν έχουμε κανέναν από το ΕΛΚ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, βεβαίω έχουμε κάποιον από το ΕΛΚΑ. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Well, uh, Mr. President, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει επιστολή ε, την οποία υπογράφουν οι πρόεδροι Μορέρα και Μπροκ και η οποία συζητήθηκε στην ΑΦΕΤΑ. Όμως, θα ήθελα να ζητήσω ερμηνευτική αποσαφήνιση σχετικά με την ε, δεύτερη παράγραφο όπου αναφέρεται ότι, ε, δεν θα, ότι πρέπει να δοθούν διασφαλίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ότι τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 του πρωτοκόλου δεν θα, δεν θα έρθουν σε αντίθεση με όλα τα προηγουμένως συμφωνηθέντα. Αναφέρεται λοιπόν η έκφραση legally binding ε, νομικά δεσμευτικά από νομική απόψης. Τι εννοούμε legally binding. Βεβαίως, υπάρχει ήδη συμφωνία σύνδεσης με, την, ε, ε, με το Ισραήλ και μέσω αυτής της συμφωνίας λαμβάνουν χώρα οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Ισραήλ. Και υπάρχει και σιωπηρή συμφωνία ε, καθώς επίσης και συγκεκριμένος μηχανισμός βάσει των οποίων οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ελέγξουν τα προϊόντα τα οποία ε, προέρχονται από τα κατεχόμενα ε, ή από τα προσαρτημένα ε, εδάφη τα οποία δεν αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, αυτή η συμφωνία θα πρέπει να ε, εφαρμοστεί, να ισχύσει και σε αυτή την περίπτωση. Τι εννοούμε όμως όταν λέμε legally binding. Ε, σημαίνει ότι εάν διαστανθούμε ότι αυτή η υποχρέωση εδώ δεν καλύπτεται θα πάμε στα δικαστήρια. Ε, θεωρώ ότι χρειάζεται περαιτέρω αποσαφήνιση του σημείου αυτού, έτσι ώστε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Thank you. Um, um... Ευχαριστούμε. Σοσιαλιστές, εσείς έχετε κάποιον που θέλει να λάβει τον λόγο. Εσείς, καλώς ήρθατε. Έγκαιρα φτάσατε. Um, on the, um, CAA για το CIA. Ακούμε τα σχόλια των ομάδων παρακαλώ. Θα θέλατε να προχωρήσω στους φιλελεύθερους και μετά να επανέλθω σε εσά. Yes, uh, <clears throat> Σας ευχαριστώ. Εχθές κιόλας είχαμε μια συμβιβαστική, ας το πω έτσι, τοποθέτηση που διαπραγματευτήκαμε. Και αυτή η ερώτηση θα διανεμηθεί αντίστοιχα για να την έχετε. Θέλουμε πράγματι δεσμευτικό, ένα δεσμευτικό σύστημα να θεσμοθετηθεί και γι' αυτό θα θέλαμε το legally binding, νομοθετικά δεσμευτικό, νομικά δεσμευτικό να ενταχθεί εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Um, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ομάδα μας ήταν υπέρ να καταλήξουμε σε ψήφιση και έγκριση. Παρότι κατανοούμε βέβαια ότι υπάρχουν κάποια ερωτηματικά που απομένουν και θα έπρεπε και να απαντηθούν. Και συμμετείχαμε και στην, ε, στις ερωτήσεις, στη διατύπωση των ερωτήσεων αυτών. Ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή πραγματικά ανησυχούμε για τις καθυστερήσεις. Διερωτόμαστε πώς εξυπηρετεί την αξιοπιστία το κύρος ε, του Ευρωκοινοβουλίου και της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής. Ε, κατανοώ τα θέματα που αφορούν δραστηριότητε και τεχνικού χαρακτήρα θέματα, όμως είναι κάτι αποθαρρυντικό αυτός ο βραδύς ρυθμός για τα θέματα τα που αφορούν τη διεργασία, τη διαδικασία. Εσείς εξ ονόματος των Πρασίνων παρακαλώ, ευχαριστώ. Μας ικανοποιεί ο συμβιβασμός που επετέφθη. Ρωτήσατε σε σχέση με το νομικά δεσμευτικό τι είναι. Είναι στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου η νομική αυτή δέσμευση. Το θέμα είναι ποιες είναι οι διασφαλίσεις αυτές για τη νομική δέσμευση, διότι τι μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κοινοβούλιο ως ε, εχέγγυα και όσον αφορά δέσμευση, δέσμευση ως προς τι και με ποιο χαρακτήρα και θα πρέπει και αυτό να αποσαφινιστεί έτσι. Δηλαδή, απλώς μόνο δεσμευτικού, δεσμευτικού χαρακτήρα ή δεσμευτικά δεν ε, το επεξηγεί. Και σε σχέση με τον ε, συμβιβασμό θα θέλαμε να ξανανοίξει η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για να μπορέσει να τροποποιηθεί για τα θέματα της ε, νομικής δέσμευσης. Μας ικανοποιεί όμως ο συμβιβασμός που επετεύχθη. Εσείς να επανέλθετε πολύ σύντομα. Δεν καθυστερούμε τη διαδικασία αυτή, εντάξει. Βήμα προς βήμα πρέπει να υπάρξει εδώ αυτή η ρύθμιση, η προσέγγιση των όρων και προϋποθέσεων. Όταν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις τηρούνται και τηρηθούν, το αργότερο τον Οκτώβριο τότε, θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε προς έγκριση Κατά τούτο λοιπόν δεν νομίζω να είναι επιβράδυνση ή καθυστέρηση των διαργασιών, των διαδικασιών, αλλά σαφείς όροι και προϋποθέσεις που θέτουμε για να διευθετηθεί το ζήτημα. Um, Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Μπέρντ. Εσείς παρακαλώ. This point was raised. Ο κ. Κασουλίδης, αυτό το σημείο εθίγει για να καταχωρηθεί στα πρακτικά ότι υπάρχει αυτό το ερωτηματικό, αυτό το ερώτημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ΕΡΚ δεν θα τηρήσει το συμβιβασμό και δεν σημαίνει ότι το ΕΡΚ δεν θα υπερψηφίσει του να αποσταλεί αυτή η επιστολή με αυτόν τον τρόπο. Well, e Ευχαριστώ. Η θέση των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών είναι να, ευχαριστήσουμε, να, ευχαριστηθούν, να ευχαριστήσουμε όλους για την συνεργασία και το επικοδομητικό πνεύμα με το οποίο αυτή η προφορική ερώτηση συντάχθηκε. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα με την παράγραφο 1. Δεν είμαστε κατά της προφορικής ερώτησης σε σχέση με την ψηφοφορία. Αν ετίθετο προς ψηφοφορία θα μπορούσαμε να απέχουμε. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα το οποίο αναφέρθηκε πιο πριν. Να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θέση της. Όλοι οι άλλοι ε, εξέφρασαν τι απόψει του. Η Γκουε, η Ενωτική Αριστερά, συγγνώμη που σα ξέχασα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματο τη ε, Ενωτική Αριστερά και των Βόρειων Πρασίνων τη Σκανδιναβία, θέλουμε να πούμε ότι συμμεριζόμαστε αυτό το συμβιβασμό και σε σχέση και με την προφορική ερώτηση για τη συζήτηση που έχουμε γι' αυτό το θέμα θα έλεγα μάλιστα χρειαζόμαστε μεγαλύτερη σαφήνεια για τα θέματα που είναι νομικά δεσμευτικά και θα θέλαμε πραγματικά να κάνουμε την προσπάθεια να αποσαφηνίσουμε γιατί πράγμα γίνεται λόγος εδώ αντί να πούμε ότι υπάρχει και δημιουργείται μια άλλη φαιά ζώνη εδώ μια ζώνη αβεβαιότητας. Προ όφελο του να επιληθεί το θέμα, νομίζω ότι αυτή η ερώτηση μπορεί να συνεισφέρει θετικά. Πρόεδρος, ρωτούσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν ήθελε να σχολιάσει ακριβώς πιο πριν και να μας δώσει κάποιες ε, απόψεις για το ποια είναι η δική της προσέγγιση σε αυτό το θέμα, για την, ε, το ζήτημα του νομικά δεσμευτικού χαρακτήρα, legally, binding. Ο κύριος Μόντ, όχι, ο κύριος Μόνος, το συγγνώμη, παρακαλώ. Um, I, think it's Η κυρία Μούνιος μάλλον και όχι μόνος, μάλιστα. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη φάση θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφουγκράστηκε, άκουσε προσεκτικά όλα τα σχόλιά σας και ουσιαστικά λάβαμε την προφορική ερώτηση και είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι να απαντήσουμε στην ε, σύγκληση της Ολομέλειας στην Ολομέλεια. Δεν νομίζω ότι είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα να αποσαφηνίσει αυτό το ζήτημα εδώ και τώρα όπως προτείνεται σε μια προφορική ερώτηση θα προτιμούσαμε να τηρήσουμε τη θέση μας την οποία θα την παρουσιάζαμε στην απάντησή μας στην Ολομέλεια όσον αφορά την προφορική αυτή ερώτηση. Εντάξει αυτό για τα πρακτικά θα ψηφίσουμε προς έγκριση αύριο για αυτή την ερώτηση. Ο κύριος Γκάρερ παρακαλώ. Συγγνώμη όμως ζήτησα εγώ. Δεν θα ήταν δυνατό να υπάρξει ένα συμβιβασμός που θα γινόταν δεκτός και έτσι θα μπορούσαμε σε σχέση με την ξεχωριστή ψηφοφορία για την παράγραφο που ζητήσαμε να υπάρξει μια αποσαφήνιση του δεσμευτικού χαρακτήρα. Θα μπορούσε να γίνει αυτό, όχι, σε σχέση με το, την πρόταση του συμβιβασμού. Υπάρχει τέτοια πρόταση για το νομικό, νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα. Το ΕΛΚ είναι κατά του να υπάρξει ο νομικά δεσμευτικός χαρακτήρας ή όχι. Μπορείτε να αποσαφηνίσετε τη διαδικασία. Ποια είναι πρόεδρε αν δεν υπάρχει συμβιβασμό σχετικά με αυτό, κάποιο συμβιβασμό, θα θέλαμε να ψηφίσουμε. Το να μιλήσει για λογαριασμό του. Αλλά δεν υπάρχει νομίζω κάποια άλλη αντίσταση. Ο κύριος Κασουλίδης, πρόεδρε, δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω παρά να επαναλάβω αυτά τα οποία είπα πιο πριν, ότι εμεί θα ψηφίσουμε υπέρ. Δεν θα είμαστε κατά τη δια, legally, νομικά, δεσμευτικά δεσμευτικού χαρακτήρα. Θέλουμε να καταχωρηθεί αυτό στα πρακτικά ως παρατήρηση και θα δούμε ποια θα είναι τα περαιτέρω βήματα και διαβήματα σε αυτή τη διεργασία και θα κρίνουμε ποια θα είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ολομέλεια για αυτό το θέμα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα διαρρήξει το συμβιβασμό και θα τον ακυρώσει. Εμείς παραμένουμε στη συμφωνία που επιτεύχθηκε. Πρόεδρος, υπάρχει λοιπόν ένα συμβασμός από ό,τι γνωρίζω για αυτό το θέμα και θα ψηφίσουμε αύριο σχετικά. Εντάξει, συμφωνείτε πολύ καλά. Ο Μπέρντ είναι εδώ παρόν. Και παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο. Α, Μπέρντ, συγγνώμη. Να επανέλθουμε στο δικό σου θέμα. Σε κάποια λεπτά θα πρέπει να αποχωρήσω και ο Ντέβιτ θα, είναι θα αναλάβει την Προεδρία. Ζητώ συγγνώμη. Η αντιπροσωπεία, ad hoc αντιπροσωπεία στην Κολομβία και το Περού. Κάποια σχόλια μπορείς να μας δώσεις και να μας πει την άποψή σου για τα ε, σχετικά θέματα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα υπάρξει και γραπτή έκθεση που θα, θα κατατεθεί και κατά τη σύνοδο του Ιουλίου σύντομα θα μπορέσουμε να τα δούμε αυτά. Όλοι θα έχετε την ευκαιρία να έχετε διαβάσει και τη γραπτή έκθεσή μας. Θεώρησα ότι ήταν αναγκαίο όμως έτσι άμεσα να σας ενημερώσω μια αντιπροσωπεία λοιπόν από πλευρά μα πήγε στην Κολομβία και το Περού. Πολύ σύντομη διάρκεια. Μία μέρα στο Περού, μία μέρα στην Κολομβία περάσαμε. Και το ψήφισμα που στην κοινοβουλευτική μα επιτροπή εγκρίναμε και που και στην Ολομέλεια εγκρίθηκε <clears throat> αφορά και τις, ε, τις κυβερνήσεις της Κολομβίας και του Περού που έπρεπε να ε, λάβουν υπόψη αυτό ήταν πολύ πιεστικό το χρονοδιάγραμμα. Είχαμε επαφές και συζητήσεις με τους δύο υπουργούς εμπορίου, Κολομβιανό και Περουβιανό. Περουβιανό. Είχαμε και συζητήσεις με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών στην Κολομβία και το Περού, με εκπροσώπους των επιχειρηματικών κύκλων και βιομηχανικών κύκλων και στην Κολομβία και στο Περού. Συζητήσεις επίσης με τα κοινοβούλια και στο Περού και στην Κολομβία και εκπροσώπους τους και είχαμε επαφές και συζητήσεις και με την ε, αναπληρώτρια Υπουργό Εξωτερικών της Κολομβίας και τον Υπουργό Εξωτερικών του Περού. Όλα αυτά στο τέλος τέλος ε, μας οδήγησαν και με τους δύο προέδρους να έχουμε επαφή, με τον πρόεδρο Σάντος και τον κύριο πρόεδρο Ουμάλα του Περού, ο πρώτος της Κολομβίας. Και με όλες αυτές τις συζητήσεις και επαφές αγαπητοί συνάδελφοι, το ψήφισμά μας ε, ο Νταβίτ και εγώ από κοινού παρουσιάσαμε τις θέσεις μας και τα αιτήματά μας λέγοντας ότι χρειαζόμαστε ένα δεσμευτικό ε, οδικό χάρτη για την ενίσχυση των ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, του περιβάλλοντος ε, για, που θα εφαρμόζονται και θα αφορούν και την Κολομβία και το Περού. Και μπορώ να σας πω ότι από όλες αυτές τις συζητήσεις οι αντιδράσεις των εταίρων μας ήταν πολύ θετικές και επικοδομητικές. Έχουμε τη δέσμευση και των δύο κυβερνήσεων Περού και Κολομβίας, ρητά και κατηγορηματικά και των δύο προέδρων των ιδίων, ότι οι δύο αυτές κυβερνήσεις με θετικό πνεύμα θα αντιμετωπίσουν τα αιτήματά μας. Και ο κύριος πρόεδρος της Κολομβίας σαφέστατα ανέφερε και προσέθεσε ότι αυτό δεν είναι μόνο ένα συμφέρον το οποίο ικανοποιεί επειδή εμείς το διεκδικήσαμε και το απαιτήσαμε αλλά φυσικά και οι ίδιοι από τις ίδιες προσπάθειες ε, της Κολομβίας απορρέει. Η κατάσταση στην Κολομβία πρέπει με αυτόν τον τρόπο να βελτιωθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν αναγνωρίζουμε και διαπιστώνουμε ότι η αναγνώριση των μεταρρυθμίσεων, ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν ακόμα επαρκώς αντιμετωπίσει ικανοποιητικά τα προβλήματα, είναι δεδομένη αυτή η τοποθέτηση. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα αυτής της σύγκλησης. Και σε αυτή η δέσμευση των δύο προέδρων και των δύο κυβερνήσεων ελπίζουμε ότι θα συνεισφέρει ώστε σε μικρό χρονικό διάστημα και από τις δύο πλευρές να υποβληθεί ο δικός χάρτης ο δικό χάρτη πώ θα πορευτούμε στο μέλλον, που μπορούμε να το συζητήσουμε και το ένα ή άλλο θέμα να το ε, τροποποιήσουμε ή να προβάλλουμε τι δικέ μα ε, θέσει. Στο τέλος τέλος πιστεύω ότι η αντιπροσωπή αυτή ήταν πολύ ικανοποιητική όσον αφορά το αποτέλεσμά της. Είχαμε πολυάριθμους εκπροσώπους κυβερνήσεων, κοινοβουλίων και άλλων εκπροσώπων που πληροφορήθηκαν για τα δικά μας αιτήματα με αυτή μας την επίσκεψη και κατέστη σαφές ότι υπάρχει σαφής αντίδραση, θετική αντίδραση και ανταπόκριση στην οποία μπορούμε να βασιζόμαστε από το Περού και την Κολομβία. Ευχαριστώ. to... Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κέλλερ και μετά στον πρέσβη για την Κολομβία, αν θέλει να σχολιάσει. Παρακαλώ. Και περνάω και την Προεδρία ευχαριστώ για αυτή την έκθεση. Ήθελα μόνο να θέσω ένα επιπλέον ερώτημα. Το ταξίδι έγινε επειδή ε, έχουμε ακροάσει της επιτροπή. έτσι. Ποια ήταν ε, η αίσθηση των Ευρωβουλευτών για αυτή τη συμφωνία. Υπήρξε μεγάλη ικανοποίηση, υπήρξαν ε, επικρίσεις, κριτικές παρατηρήσεις. Ποιες επικρίσεις ακούστηκαν στην Κολομβία ή το Περού. Ενδιαφέρον θα ήταν να ακούγαμε αν υπήρξαν τέτοιες αντιδράσεις και από την κοινωνία των πολιτών δεν ξέρουμε ποιες ομάδες συναντήσατε. Ποια ήταν εκεί η αίσθηση, ποια ήταν σημεία επί των οποίων ε, ασκήθηκε κάποια κριτική ή επικρίσεις. Ποια ήταν η δική τους αντίδραση σε σχέση με το ότι σε μικρό χρονικό διάστημα θα υπάρξει αυτός ο οδικό ε, χάρτης. Ποιο είναι, πόσο είναι αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Ένας μήνας, το επόμενο έτος, κατά το επόμενο έτος. Τι γίνεται σχετικά. Ευχαριστώ. Good morning everybody. Καλημέρα σας. Ο Χέλμοντ, ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα είχα δύο ερωτήσεις που θα ήθελα εδώ να ενταχθούν. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Και είχαμε και την πρόσκληση των δύο κοινοβουλίων ε, να ε, τους επισκεφθούμε θα με ενδιέφερε για την κοινωνία αυτή των πολιτών. Ποιους εκπροσώπους, ποιοι εκπρόσωποι ήταν αυτοί που εκπροσωπήθηκαν και συμμετείχαν ιδιαίτερα εδώ σε σχέση με τις ε, ακροάσεις που έχουμε πολλές φορές ε, ε, συζητήσει για τις τοποθετήσεις για το ψήφισμά μας ήταν άμεσα εκπρόσωποι των θυμάτων των οικογενειών ή οικοί των θυμάτων ή άλλων που είχαν ας το πω έτσι την εντολή να συμμετάσχουν σε σχέση και με τους ηθαγενείς πληθυσμούς και εκπροσώπους τους υπήρξε δυνατότητα τέτοια τοποθέτηση ε, για αυτή τη συμφωνία ή όχι. Και δεύτερον για τον οδικό χάρτη που αναφέρατε και πρόσεξα, έχουμε δύο εξελίξεις ε, αυτή την εβδομάδα. Αφενός είπα τον πρώην ε, στρατηγό Σάντος και τον πρόεδρο Ουρίμπε ε, απευθύνθηκε, κατηγορίες για την δραστήρια ε, ενεργό συμμετοχή τους σε δολοφονίες ε, και με εκπροσώπους και συμμετοχή της μαφίας, ε, συμμοριών. Θα με ενδιέφερε υπήρξε κάποια τέτοια αναφορά ή συμμετοχή και για τους εκπροσώπους των θυμάτων της κοινωνίας των πολιτών. Υπάρχει, υπήρξε κάποια τέτοια αντίδραση και για να επανέλθω στην τοποθέτηση όσον αφορά τον στρατηγό, την κατάσταση του με την ε, εισαγγελία στο Περού και την ε, Κολομβία. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο είχαμε επισκέπτες που μας ε, επέστησαν την προσοχή ότι στις ανακρίσεις θα πρέπει να υπάρξει η διακρύβωση του λόγου των δολοφονιών αυτών των συνδικαλιστών και πρέπει να αποσαφινιστούν όλοι αυτοί οι λόγοι για τους δολοφονημένους αυτούς ε, από πλευρά των συνδικάτων των εργαζομένων. Και θα πρέπει και αυτό να δούμε αν διαδραματίζει ή διαδραμάτισε ένα ρόλο σε αυτές τις επαφές. Ευχαριστώ. Κύριε Πρέσβη, θέλετε να αντιδράσετε κι εσείς στις ερωτήσεις, στις παρεμβάσεις που ακούστηκαν. Όχι. Καλώς. Μπέρτ τότε. Εσείς. Φυσικά θέλω να τοποθετηθώ. Ναι, λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, στις συζητήσεις στα κοινοβούλια οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις δεν είχαν εκπροσωπηθεί. Όμως με τις ΜΚΟ είχαμε ξεχωριστές επαφές και συζητήσεις. Στην Κολομβία την ίδια με το συνολικό φάσμα, το σύνολο του εύρους των εκπροσώπων ακριβώς ε, υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, ε, ένα ευρύτατο φάσμα οργανώσεων και εκπροσώπων τους ήταν παρόντες και εκπροσωπήθηκαν, με εξαίρεση τους, τα συνδικάτα, ιδιαίτερα της ΚΟΥΤ αυτό ίσως ε, εξηγείται, επεξηγείται και συνεχίζει το ερώτημα της κυρίας Κέλλα σαν προοπτική ότι φυσικά στην Κολομβία η έγκριση για αυτή τη συμφωνία είναι πολύ μεγάλη η θετική προσέγγιση. Θα έλεγα και πάνω από 90% ε, των πολιτικά ε, αρμόδιων είναι θετικά διακείμενοι έχουμε το ε, ε, διαφορές σε σχέση με το κόμμα Πόλο και σε συζητήσεις ε, που είχαμε, για, ακόμα και κάποιοι από αυτούς είναι σε, σε σχέση με αυτή τη συμφωνία υπέρ. Κατά τούτο η αντίδραση στο Κοινοβούλιο ήταν κάπως ευθυγραμμισμένη στη δική μας γραμμή, ότι πρέπει δηλαδή να υποστηριχθεί αυτός ο δικός χάρτης σε σχέση με την τοποθέτηση ότι δεν χρειάζεται ο δικός τέτοιο χάρτη και απλά και μόνο πρέπει να προσυπογραφεί η συμφωνία. Έτσι λοιπόν η αντίδραση, η τοποθέτηση συνολικά ήταν μάλλον υποστηρικτική σε σχέση με τις προσπάθειές μας και τα αιτήματά μας από την κοινωνία των πολιτών. Μεγάλη συνένεση ε, σημειώθηκε να κινηθούμε με αυτόν τον τρόπο για την συμφωνία αυτή. Και τώρα, στη συνέχεια, συζήτησα εκ των υστέρων με τις τρεις ε, οργανώσεις συνδικάτων στην Κολομβία. Υπάρχουν για λόγους αρχής κάποια επιχειρήματα που τους κάνουν να απορρίπτουν αυτή τη συμφωνία. Για πολιτικούς λόγους, ότι το ελεύθερο εμπόριο σε αυτά τα πλαίσια δεν είναι το ορθό, το σωστό για εκείνους. Δεν είναι αυτό η δική μου θέση, αλλά πρέπει να το δεχτούμε αυτό ότι είναι η δική τους θέση και να το σεβαστούμε. Γι' αυτό θα πρέπει να σε σχέση με την ανταπόκριση στα δικά μας αιτήματα ήταν μάλλον πολύ συγκρατημένη από τα συνδικάτα. Όμως συνολικά υπάρχει, θα έλεγα, καλοδεχούμενη, ε, είναι ευκταία και με συνένεση γίνεται δεκτή αυτή η πρόταση από την κοινωνία των πολιτών. Είχαμε και ένα σεμινάριο σε πανεπιστημιακό επίπεδο που από τους πιο διαφορετικούς εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών συμμετείχαν εκπρόσωποι. Και έτσι και στο Περού δεν είδα κάποια φωνή να γύρεται εναντίον, κάποια διαφωνία κατά αυτής της συμφωνίας. Ούτε όμως και κατά του δικού μας αιτήματο να υπάρξει ένας οδικός χάρτης για τη μελλοντική μας πορεία. Πιστεύω ότι στο Περού η έγκριση για αυτή την εμπορική συμφωνία είναι ακόμα μεγαλύτερη από τη έγκριση και η συνένεση στην Κολομβία. Αυτή είναι η προσωπική μου εντύπωση για έναν τομέα του Περού που έχει προβλήματα είναι ο γαλακτοκομικός τομέας. Είναι ο φόβος εισαγωγών για γαλακτοκομικά προϊόντα από την Ευρώπη που τους κάνει να διαφωνούν. Και αυτό την κυβέρνηση στο Περού, η κυβέρνηση στο Περού το αναγνώρισε και το έλαβε υπόψη και για τα γαλακτοκομικά προϊόντα θα υπάρξουν μεγαλύτερες προθεσμίες ε, σε σχέση ίσως με τη συμφωνία αυτή. Και το τελευταίο σε σχέση με την ε, εκπνοή θα είναι την προθεσμία για εκπνοή της συμφωνίας 17 χρόνια μετά από αυτή την ε, ας χρονική στιγμή έναρξης. Θα εισαχθούν μέτρα λοιπόν ώστε ο γαλακτοκομικός τομέας και οι μικροί ε, κτηνοτρόφοι, μικροκτηνοτρόφοι να μην πληγούν λόγω εισαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων σε αυτές τις χώρες. Εξαγωγές δηλαδή από την Ευρώπη προς τις χώρες Λατινικής Αμερικής και τα θέματα, για τα θέματα δικαιοσύνης. Και στην η Κολομβία είχαμε επαφή με εκπροσώπους της εισαγγελίας και στο Στρασβούργο με τον Γενικό Εισαγγελέα που εδώ και δύο μήνες έχει αναλάβει αυτό το αξίωμα αυτές τις αρμοδιότητες. Υπάρχουν πολλές προσπάθειες που καταβάλλονται από πλευράς της Γενικής Εισαγγελίας να διακριβωθούν αυτά τα γεγονότα και να φωτιστεί τι έγινε. Και οριζόντια, εγκάρσια να μπορέσουν να γίνουν ε, διακριβώσεις και εξετάσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις διαφορετικοί τομείς της Γενικής Εισαγγελίας ε, κάνουν παράλληλες διακριβώσει, διότι δεν υπάρχει αυτό το οριζόντιο εγκάρσιο επίπεδο συμμετοχής όλων προς μια κοινή κατεύθυνση. Και όσον αφορά τους, ε, τα, θέματα συνδικαλιστών και εργαζομένων, ένα ειδικό τμήμα ε, πρόκειται να επιληφθεί αυτών των ε, ερευνών από τη Γενική Εισαγγελία. Όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων από την κυβέρνηση. Πρέπει όμως όλα αυτά να διασφαλιστούν με ένα δεσμευτικό δικό χάρτη και να δούμε πότε ποια βήματα και πράξεις και ενέργειες θα διασφαλίζονται διότι είχαμε και μια έκθεση για την ατιμορρησία στην Κολομβία που δημοσιεύθηκε, δημοσιοποιήθηκε και διαπιστώνεται ότι υπάρχουν 1500 τέτοιες περιπτώσεις βίας, έκδηλης βίας και βιοπραγιών κατά εκπροσώπων των εργαζομένων συνδικαλιστών που δεν έχουν διακριβωθεί και εξεταστεί σε βάθος από τις αρχές. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει με ένα νέο σύστημα διακριβώσεων και εξετάσεων να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν τεράστια βουνά, στίβες φακέλων και θα έλεγα ε, χαρτοφυλακίων ε, για όλες αυτές τις περιπτώσεις, για όλα αυτά τα θέματα. Πρέπει όλα αυτά να ε, εξεταστούν σε βάθος. Δεν είναι δυνατόν να αφαιθούν αυτές οι περιπτώσεις αδιακρίβωτες. Ε, και γι' αυτό η εντύπωσή μου είναι ότι κάτι κινείται τώρα, κάτι έχει αρχίσει να κινητοποιείται. Πρέπει όμως ε, να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει συνέχεια και να παρακολουθήσουμε αυτή τη διεργασία. Ε. Ευχαριστούμε. Την επόμενη εβδομάδα νομίζω θα είναι διαθέσιμη έκθεση και θα μοιραστεί ως πρέπει. Σημείο 7 στην ημερήσια διάταξη τώρα πρόκειται για την επέκταση ε, διατάξεων Συμφωνίας τελικής Σχέσης και Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουσβεκιστάν στο διμερές εμπόριο κλωστοφαντευτικών ε, προϊόντων. Η συγγητής είναι ο Ζόρζο Σαμπίν Κούτας. Η ΙΝΤΑ έχει ήδη εγκρίνει μια προσωρινή έκθεση για το θέμα αυτό και η ιδέα ήταν να βασιστούμε στην ε, διαδικασία που προβλέπεται βάσει του άρθρου 81, παράγραφος 3, όσον αφορά το εμπόριο παιδιών, βασικά την χρήση παιδιών σε αυτό το εμπόριο. Υπήρξε σύσταση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή και η Ολομέλεια, όπως γνωρίζετε, συμφώνησε με τις προτάσεις της ΙΝΤΑ ε, η διαδικασία βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί και η ίντα πρέπει να δώσει συνέχεια. Ο πρόεδρος της ίντα έστειλε επιστολή στην Επιτροπή και το Συμβούλιο για την συνάντηση αυτή. Ο κύριος Δεβίν είναι εδώ, έτσι. Πρόεδρε, ο κύριος ε, Κισό είναι στο δρόμο. Έρχεται. Καλώς, έτσι καλώς δεν θα μιλήσει πρώτος. Και εκ μέρους του Συμβουλίου Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ο κύριος Μαλντονάντο. Είναι εδώ. Ε? Είναι, είναι. Ωραία. Καλώς. Συνεπώς, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας πρώτα απ' όλα, τον Ζόρζ Σαμπίν Κούτας, να μας πει πού βρισκόμαστε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτον, Θέλω να σας υπενθυμίσω, πέρα από αυτήν την προσωρινή έκθεση, στην οποία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος μας, να σας πω ότι το Κοινοβούλιο μας ζήτησε να εγκρίνουμε την διεύρυνση της Συμφωνίας εταιρική Σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του Σπικιστάν, όσον αφορά το εμπόριο κλωστεφαντουργικών προϊόντων. Έχουμε ακούσει ότι χρησιμοποιούνται τα παιδιά σε καταναγκαστικά έργα. Εκεί, καταναγκαστική εργασία. Στο βαμβάκι λοιπά. Στον ε, τομέα αυτών των κλωστοφαντουργικών λοιπόν και αποφασίστηκε να αναβάλουμε τη συμφωνία του πρωτόκολλου προκειμένου η Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις δικές μας συστάσεις. Και αυτές ακριβώς θέλω να σας υπενθυμίσω. Πρώτον, αυτό που ζητάμε είναι Το Συμβούλιο και η Επιτροπή να ζητήσουν από το Σουμπεκιστάν να δεχτεί τριμερή αντιπροσωπεία παρατηρητών για να δούμε αν μπορούμε να ελέγξουμε και την κατάσταση με ελευθερία βέβαια διακίνησης εκεί. Να δούμε δηλαδή τι γίνεται όταν μαζεύουν τον μπαμπάκι στη χώρα αυτή και να εκτιμήσουμε έτσι το κατά πόσο τηρείται το πρωτόκολλο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Αυτό ζητήσαμε. Θέλουμε να αναλυθεί η δυνατότητα αυτή, να ερευνήσουμε την κατάσταση και όσον αφορά τις προτιμησιακές συμφωνίες. Θέλουμε επίσης να αναλύσουμε μια νομοθετική πρόταση για να υπάρχει ένας μηχανισμός αποτελεσματικός όσον αφορά την ιχνηλεσιμότητα των προϊόντων των κλωστιφαντουργικών για να δούμε αν όντω χρησιμοποιούνται παιδιά στη δουλειά αυτή όχι. Ζητούμε από τις αρχές του Ουσβεκιστάν να τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Ουσβεκιστάν έτσι κι αλλιώς έχει υποστηρίξει ήδη και έχει υπογράψει διάφορες συμφωνίες για την απαγόρευση της παιδικής εργασίας κτλ. Παρ' όλα αυτά, στην πράξη δεν φαίνεται όλα αυτά να ισχύουν. Συνεπώς, αυτή ακριβώ είναι και η ερώτησή μου. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Σπικιστάν και κατά πόσο υπάρχουν πραγματικές δυνατότητες στο φθινόπωρο όταν αρχίζει η συλλογή του βαμβακιού, αν μπορούμε να οργανώσουμε μια τέτοια αντιπροσωπεία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας στο Ουσβεκιστάν. Σε τι βαθμό η Επιτροπή επίσης στηρεί τις συστάσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά την ε, έρευνα αυτή που ζητάμε για την αναστολή των προτιμήσεων του σίγμα και τι κάνει για τον μηχανισμό αυτό λεσιμότητας ε, που ζητάμε ώστε να ξέρουμε κατά πόσο χρησιμοποιείται καταναγκαστική παιδική εργασία ή όχι. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Νομίζω είναι σαφής η ερωτήση Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή, την Επιτροπή σας που μας δίνει την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε το θέμα από τη δικιά μας την πλευρά. Είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα. Σας υποσχεθήκαμε σε αυτήν την ίδια αίθουσα να δράσουμε έτσι ώστε να εξηγήσουμε στο Ουσβικιστάν ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέραν της συνεργασίας με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Επίσης, υποσχεθήκαμε ότι θα πιέσουμε περισσότερο τη χώρα, κάτι το οποίο κάναμε. Οι διπλωματικές μας προσπάθειες οδήγησαν στην αναγκαιότητα να καταλάβει το Ουσβεκιστάν ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση πέρα τη συνεργασία αυτής. Τον Νοέμβριο τώρα που μας πέρασε, οι υπηρεσίε τη Επιτροπή στην Τασκένδη οργάνωσαν μία αποστολή μαζί με την Υπηρεσία εξωτερική δράση. Είχαμε διαβουλεύσει, με τους εκπροσώπους του Εθνικού Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Σπίκιστάν, με την Αντιπρόεδρο του Υπουργείου Εργασίας, αλλά και με εκπροσώπους και της UNICEF και, της, ε, και του Γραφείου Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Το μήνυμα που περάσαμε στο Ουσβικιστάν, ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από τη συνεργασία με το Εθνές Γραφείο Εργασίας, κάτι το οποίο επαναλάβαμε ξανά και ξανά και στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκή Ένωσης και του Ουσβεκιστάν. Και το Συμβούλιο αυτό είναι η θεσμική ετήσια συνάντηση που έχουμε, η πιο σημαντική δηλαδή, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ουσβεκιστάν. Στη συνέχεια υπήρξαν ε, και άλλες επαφές που οργάνωσε ο πρέσβης μας εκεί επιτόπου, αλλά συναντηθήκαμε και με τον πρέσβη του Σμπικιστάν εδώ στις Βρυξέλλες. Είχαμε τακτικές συναντήσεις επίσης και με τον ειδικό σύμβουλο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας εδώ στις Βρυξέλλες. Πού οδήγησαν όλα αυτά. <clears throat> Το Ουσβεκιστάν αποφάσισε στα πλαίσια μιας θεσμικής συνάντησης που είχαμε όσον αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις, αποφάσισε λοιπόν να οργανώσει μία διάσκεψη για την εφαρμογή των ε, συμφωνιών του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και ιδιαίτερα όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών. Η διάσκεψη αυτή έλαβε χώρα στη Δασκένδη, στις 3 Μαΐου που μας πέρασε. Συμμετείχαν σε αυτήν και Διεθνή Οργανισμό Εργασία και υπηρεσίε τη Επιτροπή αλλά και οι υπηρεσίε τη εξωτερική δράση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το Σουβεκιστάν πήρε πολύ στα σοβαρά την οργάνωση αυτής της συνάντησης. Η Επιτροπή από την πλευρά της έπαιξε ένα ρόλο διαμεσολαβητή. Προσπάθησε να διευκολύνει το διάλογο αυτό και κατά τη διάρκεια της διάσκεψης αυτής καθ' αυτής, αλλά και κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων συναντήσεων που έγιναν, κυρίως σε υπουργικό επίπεδο. Συνεισφέραμε λοιπόν, πιστεύω, να ξεκινήσει ένας νέος δρόμος επαφών ανάμεσα στο Ουσβεκιστάν και το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. Το μήνυμα ήταν το ίδιο. Χρειάζεται αποτελεσματική πραγματική συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. Τι σημαίνει αυτό τώρα συγκεκριμένα και για να απαντήσω και στις ερωτήσεις σας. Το Ουσβεκιστάν σημαίνει ότι πρέπει να δεχτεί μία αποστολή ελέγχου επιτόπου. Πολύ πρόσφατα το Ουσβεκιστάν στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε την ε, βούληση του Ουσβεκιστάν να συνεργαστεί με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την Σύμβαση 138 που μιλάει για τις προδιαγραφές ε, εργασίας και μια άλλη που μιλάει για τα δικαιώματα των παιδιών. Κάθε τέτοια συνεργασία βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να μπορούμε και να επαληθεύσουμε ότι στην πράξη εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά. Η Επιτροπή λοιπόν παρακολούθησε και την ε, ετήσια διάσκεψη του Διεθνής Οργανισμού Εργασίας από το Μάιο μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Φέτος η διάσκεψη αυτή δεν κατέληξε σε κανένα συμπέρασμα από την Δικευμένη Επιτροπή του για την παιδική εργασία και ιδιαίτερα για το Σβεκιστάν. Δηλαδή η Επιτροπή, μάλλον η ομάδα αυτή, δεν ε, ανέφερε προβλήματα με την παιδική εργασία στο Σβεκιστάν. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή ανάμεσα σε άλλες δράσεις της καθόρισε και ένα πρόγραμμα αρρωγής στις γεωργικές μεταρρυθμίσεις του Σπικιστάν. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η γεωργία και η μεταρρύθμιση της γεωργίας ε, μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην κατάργηση της παιδικής εργασίας. Το πρόγραμμα αυτό συνεχίζεται και φέτος και πρόκειται για 10 δισεκατομμύρια ε, ευρώ. Πολύ σημαντικό δηλαδή. Πριν λοιπόν απαντήσω στη συγκεκριμένη ερώτηση που κάνατε Θέλω να σας πω ότι εμεί πιστεύουμε ότι το Ουσβεκιστάν έκανε πραγματικές προσπάθειες τους τελευταίους έξι μήνες και ανταποκρίθηκε στην πίεση που δέχτηκε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την εκθεσή του, αλλά και από την ε, Κομισιόν. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι είναι ζωτική σημασία στο εξή. Το Ουσβεκιστάν έστειλε ένα μήνυμα στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας στη Γενέβη λέγοντας ότι δέχεται τελικά την αποστολή αυτή αξιολόγησης η οποία θέλουμε να γίνει την ε, επόμενη περίοδο συγκομιδής ε, Βάβακος. Η αρχή δηλαδή έχει γίνει δεκτή, οπότε τώρα εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να δούμε με ποιο τρόπο θα λάβει η χώρα ακριβώς η αποστολή αυτή, για να είναι και αποτελεσματική. Το τελευταίο που θέλω να απαντήσω είναι αυτό που είπατε για τις γενικευμένες προτιμήσεις. Ξέρετε πώς δουλεύει το σύστημα αυτό η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει ε, δράσεις, έρευνας ή και να αποσύρει ε, κάτι, αλλά στα πλαίσια μιας σαφούς έκθεσης από πλευράς του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Η Επιτροπή δηλαδή βάσει των υποχρεώσεων της δεν μπορεί να καταλήξει σε μια τέτοια δράση, αν προηγουμένως το Διεθνές, ε, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας δεν πει ότι υπάρχει πρόβλημα με την παιδική εργασία, κάτι το οποίο δεν έγινε στην ετήσια ε, συνεδρίασή του. Συνεπώς νομικά δεν έχουμε στοιχεία στη διάθεσή μα για να ξεκινήσουμε μια τέτοια διαδικασία, η οποία, όπω σα είπα, βασίζεται στο γεγονό ότι υπάρχει συστηματική παραβίαση τη σύμβαση ε, του ΔΟ για την παιδική εργασία. Εκεί βρισκόμαστε, Πρόεδρε. Άρα, η αρχή για μια τέτοια αποστολή έχει κατοχυρωθεί και άρα καρποφόρησαν οι προσπάθειες τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλώ τώρα από πλευρά τη Υπηρεσία Εξωτερικών Δράση, ο κύριο Μαντονάλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά που ήδη ο κύριος Κουτσόν είπε. Ε, ως εκπρόσωπο της Επιτροπής. Συμφωνούμε απολύτως με την προσέγγιση ε, και έχουμε δουλέψει ε, πολύ στενά συνεργαστεί με την Κομισιόν καθώς επίσης και με την Δενική Προεδρία αλλά και με την Αντιπροσωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Γενέβη. Κοινή εργασία λοιπόν, τα αποτελέσματα της οποίας μας χαροποιούν. Έχουμε κοινό στόχο και με κοινή προσπάθεια προσπάθεια μπορούμε να επιτύχουμε τους επιδιωκόμενους στόχους ε, σε, συν, ε, σε αγαστή συνεργασία με την αφορόμενη χώρα, εν προκειμένου του Ουσμπικιστάν. Deployment of monitoring mission for the next... ε, για την επόμενη συγκομιδή Βαμβακιού ε, θα υπάρξει κάποια διερευνητική ε, αποστολή για να δούμε από κοντά τα πράγματα. Να προσθέσω το εξή την 19η Ιουλίου θα έχουμε ε, συνάντηση συνεργασία με το Ουσβεκιστάν στην Τασκένδη και προτιθέμεθα να συζητήσουμε ξανά ε, το θέμα αυτό έτσι ώστε να έχουμε πιο λεπτομερή ε, γνωστοποίηση των κινήσεων που θα λάβουν χώρα αργότερα. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Βλέπω ότι εδώ η ευρωπαϊκή διπλωματία υπήρξε πολύ αποτελεσματική. Πριν δώσω το λόγο ξανά στον εισηγητή, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να περάσουμε από τον Πολ Μέρφυ, τον ε, σκιώδη εισηγητή, ίσως κάποια άλλα μέλη της Επιτροπής. Και τελικά ο συνάδελφος Κούτας ως εισηγητής ε, να κάνει τα τελικά του σχόλια ή ενδεχομένως να υποβάλει περαιτέρω ερωτήσεις ε, την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως ε, είναι ο κατάλληλος χρόνος ε, για να γίνει η συζήτηση αυτή και βάσει του ψηφίσματος. Ε, φτάνει όπου να είναι η εποχή συγκομιδή στο Ουσμπεκιστάν. Και εγώ να σας πω την αλήθεια δεν δέχομαι ότι το Ουσμπεκιστάν έκανε οποιαδήποτε πρόοδο την ε, Άνοιξη ε, είχαμε καλλιέργεια ε, βαμβακιού στην οποία χρησιμοποιήθηκε παιδική εργασία αναγκαστική υποχρεωτική εργασία επομένως εγώ δεν βλέπω να έχουν αλλάξει καθόλου τα πράγματα και οι πρακτικές εάν έχουμε τα ίδια με αυτά που είδαμε την προηγούμενη φορά τότε θα έχουμε δύο εκατομμύρια παιδιά τα οποία θα έχουν ασχοληθεί με την συγκομιδή. The commission is suggesting has taken place. Well, Εν πάση περιπτώσει, ε, όσον αφορά τη θέση της Επιτροπής σχετικά με μία αναφορά ε, των προβλημάτων ε, ε, από πλευράς του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας το Ουσμπεκιστάν διεμήνησε ότι δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί μια τέτοια διερευνητική αποστολή και βεβαίως το Κοινοβούλιο είναι σαφές στο ψήφισμά του Ιχνογραφείου γραφειου εργασιας το ουσμπεκισταν διεμηνησε οτι δεν προκειται ποτε να υπάρξει τριμερής διερευνητική αποστολή με πλήρη ελευθερία κινήσεων που θα μπορεί να επισκεφθεί οτιδήποτε το ενδιαφέρον ενδιαφέρει συμπεριλαμβανομένων και των βαμβακοκαλλιεργειών. Ε, εν πάση περιπτώσει, αλλά φαίνεται ότι το, η κυβέρνηση κατέστησε σαφέ ότι δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί ε, μια τέτοια διαρευνητική αποστολή. Εν πάση περιπτώσει, να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν ε, αυτή τό το το θέμα θα αναφερθεί και στην έκθεση προόδου για την ε, ε, Κεντρική και Ανατολική ε, Ασία. Το Συμβούλιο και οι Κομισιόν πλέον έχουν ευθύνη να κάνουν ε, ε, κάτι παραπάνω, να ασκήσουν περισσότερη πίεση ε, και να πιέσουν περισσότερο την κατάσταση, να πιέσουν έτσι ώστε να υπάρξει υψηλού επίπεδου τριμερής αντιπροσωπεία στο Ουσμπεκιστάν, γιατί διαφορετικά επιτρέπουν στο, στην κυβέρνηση να συνεχίζουν με την ίδια, την ίδια πορεία και με τον ίδιο τρόπο ε, και την προηγούμενη φορά μας ε, είχε διασφαλίσει η κυβέρνηση του Ουσμπεκιστάν ότι βεβαίως συμμορφώνονται με την ε, συνθήκη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας κτλ. Τα, τα ίδια και τα ίδια λοιπόν και αυτό είναι απαράδεκτο πλέον. Thanks. Um... Πράγματι, η πρόεδρος αυτή που αναφέρεται από την Επιτροπή, πολύ καλή υπόθεση, αλλά και αυτό πρέπει να παρακολουθηθεί ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πετύχουμε κάτι σε σχέση με αυτή την αποστολή, αυτό το εγχείρημα. Και υποστηρίζω ότι πρέπει να είναι μια αποστολή όπως είπαμε εμείς στο Κοινοβούλιο και όχι οτιδήποτε άλλο και αν ότι η κυβέρνηση του Ουσμπεκιστάν δεν θα συμφωνήσει για μια τέτοια αποστολή, έχουμε διαφορετικές πληροφορίες. Ίσως μπορείτε να αποσαφηνίσετε για ποιο είδους αποστολή μιλάτε εσείς και να δούμε τι θα γίνει με την έκθεση μετά από αυτή την υψηλού επίπεδου αποστολή και να δούμε ποια άλλα βήματα και διαβήματα θα πρέπει να κάνουμε εμείς. Ευχαριστώ. Ε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλεις να υποβάλεις κάποιο ερώτημα στην Κομισιόν και ούτως ή άλλως μετά θα σου δώσω το λόγο για να ολοκληρώσεις ε, τη συζήτηση. Μετά θέλεις ή τώρα. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια θετική προσέγγιση και χαίρομαι που ακούω ότι θα οργανωθεί μια αντιπροσωπή. Έχω όμως και εγώ επιφυλάξεις όσον αφορά την κυβέρνηση του Ουσπακιστάν. Πρόκειται πράγματι να δεχτεί αυτή την αποστολή για το φθινόπωρο. Ο χρόνος πιέζει. Γι' αυτό και θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει και πάλι το διάλογο για να επιβεβαιωθεί η στάση αυτή του Ουσβεκιστάν για την ε, αποστολή του ΔΟΕ στο Ουσβεκιστάν το φθινόπωρο. Είναι σαφές ότι τόσο εμεί όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζουμε να επιμένουμε. Η έκθεση ελπίζω να είναι θετική. Αλλά καταλαβαίνετε ότι από την άλλη μεριά ο εταίρος μας δεν είναι κάποιος με τον οποίο να μπορούμε εύκολα να έχουμε διάλογο για να βρίσκουμε λύσεις. Είναι περίπλοκη η κατάσταση. Πάντως ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε μια θετική έκθεση τελικά. Και ελπίζω επίσης ότι στο τέλος η κυβέρνηση του Ουσβεκιστάν θα καταλάβει και θα συμφωνήσει με την αποστολή αυτή. Ευχαριστώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση μετά, αν επιθυμεί. Η Κομισιόν πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι επί της αρχής συμφωνούμε όλοι. Λοιπόν, η αρχή, ε, ε, ε, ε επί της ουσίας λοιπόν υπάρχει συμφωνία όσον αφορά την αποστολή τη διερευνητική ε, παραμένουν ε, να καθοριστούν οι τυπικές λεπτομέρειες. Το γεγονός είναι ότι η κυβέρνηση του Ουσμπεκιστάν έχει αποδεχτεί μια τέτοια αποστολή. Τώρα το εάν θα είναι τριμερής και άλλου είδους τέτοιες λεπτομέρειες ακόμα ε, τελούν υποσυζήτηση να παρατηρήσω ότι αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας να βρίσκονται επί τόπου για να διαπιστώσουν την πραγματικότητα. Αυτό μας ενδιαφέρει και αυτό το έχουν αποδεχτεί. Επί της αρχής λοιπόν είναι δεδομένη η συμφωνία. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα θα σας ενημερώνουμε τακτικά. Ο κύριος Μαλτονάντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, το κύριο πρόβλημα το οποίο ανέφεραν ε, οι εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας είναι η χρήση, ε, η συμμετοχή, η χρήση ανηλίκων στη συγκομιδή βαμβακιού. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το μικρόφωνο. Ωραία. Συνεχίζω. Α, μάλλον όχι, να ξαναρχίσω. Από όσα γνωρίζουμε, ακολουθώντας ε, και τα συμπεράσματα της Αρμόδιας Επιτροπής ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας στην Γενέβη, το κυριότερο πρόβλημα στο Ουσμπεκιστάν είναι η χρήση υποχρεωτικής εργασίας παιδιών, ανηλίκων, στην συγκομιδή βαμβακιού, δηλαδή από το Σεπτέμβρη μέχρι το Νοέμβρη. Ε, φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν παιδιά και στην ε, περίοδο σποράς, αλλά αυτό ε, είτε έγινε πρώτη φορά, είτε πρώτη φορά ε, το γνωστοποιείται σε Το σημαντικό είναι η περίοδος της συγκομιδής. Όσον αφορά τώρα το είδος της αποστολής, είναι γεγονός αυτό που είπαν τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, ότι το προηγούμενο χρόνο το ψήφισμα ε, για, το, για την αποστολή ανεφέρετο σε υψηλού επίπεδου τριμερή διερευνητική αποστολή. αλλά καταλαβαίνετε υπάρχουν πολλές μορφές αποστολών. Ε, μπορεί να υπάρχει μία για να διερευνήσει τις συνθήκες εργασίας, άλλη για, την, ε, για το σημείο εφαρμογής των ε, συμβάσεων. Όσον αφορά ε, το την υψηλού επίπεδου αποστολή ε, φαίνεται ότι από το Διεθνέ Γραφείο εργασία προτιμούν μια τεχνοκρατική αποστολή η οποία θα ξεκινήσει από τι ε, τεχνικέ λεπτομέρειε και, και να ερευνήσει το κατά πόσον καλύπτονται τα προβλεπόμενα από τι συνθήκε. Εμεί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να διαμεσολαβήσουμε έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εξέβρεση λύσης. Τώρα, πώς ακριβώς και ποια μορφή θα λάβει η διερευνητική αποστολή θα πρέπει να την ε, ε, ρυθμίσει και η ε, κυβέρνηση του Ουσμπεκιστάν. Το σημαντικό για μας είναι να δούμε, να διαπιστώσουμε εάν κατά τη διάρκεια της συγκομιδής βαμβακιού χρησιμοποιείται υποχρεωτική παιδική εργασία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα για μας. Μέχρι τώρα Ε, σε όλα τα έγγραφα γίνεται αναφορά σε διερευνητική ε, αποστολή χωρίς να αποσαφηνίζεται αν πρόκειται για τεχνοκρατική ή όχι, αν πρόκειται για υψηλού επίπεδου ή λιγότερο υψηλού επίπεδου κτλ. Το σημαντικό είναι να δούμε στην, στα πλαίσια της συγκομιδής τι ακριβώς γίνεται. Πάντως, εγώ, λαμβάνοντας υπόψη και άλλα παραδείγματα του παρελθόντος, ε, μπορώ να πω ότι μονάχα οι τεχνοκράτες μπορούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει πραγματικά ε, υποχρεωτική εργασία ανηλίκων ε, στους, στα χωράφια. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ε, είναι η υπηρεσία η οποία ε, αναλαμβάνει την, τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τα προβλεπόμενα στις ε, συνθήκες. Ε, ε, πάντως, την 19η Ιουλίου θα έχουμε τη συνάντηση στην οποία αναφέρθηκα στην Τασκένδη και με τους αρμοδίους αξιωματούχους του Ουσμπεκιστάν θα δούμε ποια είναι τα βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθηθούν για την οργάνωση αυτής της διερευνητικής αποστολής. Οι όροι της αποστολής αυτής ε, θα πρέπει να έχουν αποφασιστεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου, έτσι ώστε να μπορέσει να οργανωθεί αυτή η ε, διερευνητική αποστολή έγκαιρα και σωστά. Προτείνω λοιπόν να περιμένουμε μέχρι τότε Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε ε, την ε, δυνατότητα στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας να μας ε, δώσει όλα τα στοιχεία σχετικά με τη διερευνητική αποστολή, τι περιμένουμε και τι αποτελέσματα μπορεί να έχουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπενθυμίζω ότι ο εισηγητής και η δική μας επιτροπή ε, θα αποφασίσει εάν θα ξαναρχίσει η διαδικασία ε, έγκρισης ή όχι. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. <clears throat> Πίεσε ο χρόνος και όπως είναι γνωστό, τον Ιούλιο θα μπορέσουμε να περάσουμε στις θερινές διακοπές. Μέχρι τότε κάτι πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια άλλη λύση. Ελπίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα τονίσουν το θέμα και θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο στον διάλογο με την κυβέρνηση του Ουσμπεκιστάν να περάσουν αυτές τις απόψεις και θέσεις. Όμως δεν με ικανοποιεί το χρονοδιάγραμμα. Η έκθεσή μας ήταν θέμα το οποίο εγκρίθηκε την Άνοιξη. Τώρα φτάσαμε στον Ιούλιο, Ιούνιο 2012 και τι θα γίνει με τη συνέχεια αυτών των ε, θεμάτων. Το Σεπτέμβριο θα έχουμε τη συγκομιδή, της, ε, την επόμενη συγκομιδή Βαμβακιού. Ελπίζω λοιπόν οι παρατηρητές ε, να μπορέσουν ελεύθερα να κυκλοφορούν σε αυτή τη χώρα, χωρίς προσκόμματα και περιορισμούς. Τη θέση μας την καταστήσαμε απόλυτα σαφή για αυτό το θέμα. Κατά τα άλλα όμως δεν συμφωνούμε με τη διαδικασία που ακολουθείται για αυτήν την έκθεση. Le Πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν το θέμα αυτό και των τροποποιήσεων των παρατημάτων 1 και του κανονισμού του Συμβουλίου. Και έτσι θα πρέπει για κάποιες χώρες και περιφέρειες που θα πρέπει να εξεταστούν σε σχέση με αυτό το θέμα αυτού του κανονισμού. Ο Ντέβιτ Μάρτιν δεν είχε ποτέ ασχοληθεί με τόσο ακαθόδες θέμα. Ίσως μπορεί να μας ενημερώσει για τα θέματα αυτού του χαρτοφυλακίου και έτσι να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ για την ευμενή φιλική σας αυτή η εισαγωγή, Πρόεδρε, τα φιλικά σας λόγια. Τα συζητήσαμε κάποιες φορές πιο πριν. Είναι ασυνήθιστο. Εγώ θα ήθελα να πάρουμε κάποιο χρόνο και να εξετάσουμε κάποια θέματα που αξίζουν το θέμα, την προσοχή μας. Υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις δυστυχώς και πρέπει να πω προσωπικά ότι σκλήρινα τη θέση μου, την κατέστησα πιο αυστηρή τις τελευταίες εβδομάδες για αυτά τα θέματα αυτού του χαρτοφυλακίου. Όπως είπατε, είναι η πρόταση να ολοκληρωθεί η προσέγγιση που υιοθετήθηκε από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας που επέτρεπε σε 36 χώρες να ε, υποφελούνται από προτιμησιακή προνομιακή προσέγγιση στις αγορές μας για τα προϊόντα τους η πρόταση αυτή να ολοκληρωθεί η διαδικασία είναι το ότι έχουν καταργηθεί αυτά τα ε, δασμολογικά ε, προσκόμματα και θα έχουμε χώρες ολόκληρες που θα αφαιρεθούν από αυτό τον κατάλογο και θα πρέπει να αντικατασταθούν είτε με γενικευμένες προτιμήσεις, δασμολογικές προτιμήσεις ή με τίποτα άλλο. Και νομίζω είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνονται αυτές οι προτάσεις. Πήγα και στην Κένια ως μέλος της ΑΚΕ, πήγα και στη Ζάμπια και σε σχέση και με την συνάντηση που έγινε με τους εκπροσώπους της ΑΚΕ, συζήτησα με εκπροσώπους και της Αφρικής και της Καραϊβικής και όλοι αναγνωρίζουν και βλέπουν ότι είναι μια παρεμβατική, επιθετική ε, προσέγγιση και πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το θεωρούν ως ε, εκβιασμό, ως μια προσπάθεια του να ενταχθούν σε μια ε, κατηγορία που δεν θα έχουν πλέον άλλες δυνατότητες. Επίσης, θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη και να αναφερθεί από πλευράς ο δικής μας ότι διαφορετική είναι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε σχέση με τα θέματα πρόσβασης να βρεθεί κάποια λύση. Επειδή όμως έχουμε θέματα δημόσιων προμηθειών, θέματα της Σιγκαπούρης, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι πολύ περίπλοκα αυτά τα θέματα, πολύ περίπλοκη αυτή η ε, συμφωνία. Είναι δύσκολο λοιπόν για αυτές τις χώρες να ολοκληρώσουν αυτή τη ε, διαδικασία μέσα στα τακτά πλαίσια. Θα πρέπει να τερματιστούν κάποιες ε, εσφαλμένες απόψεις και προσεγγίσεις που λένε κάποιοι ότι δεν μπορούμε να παρατείνουμε και να επεκτείνουμε διαρκώς την τελική προθεσμία εκπνοής. Δεν είχαμε ποτέ μια τέτοια προθεσμία. Είχαμε το 2007 ως τέλος ε, της εξαίρεσης, ε, του πλαισίου εξαιρέσεων και ποτέ μετά από αυτή την ημερομηνία δεν υπήρξε κάποια προθεσμία εκπνοής, καταληκτική προθεσμία. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό αλλά σε σχέση με το 2014 ως προθεσμία είναι ανέφικτο να την ε, υλοποιήσουν κάποιοι εταίροι μας. Δεν θα είναι λοιπόν μια κινητή μεταθέσιμη ημερομηνία όταν θα ε, εγκριθούν οι τροπολογίες θα υπάρξει καθορισμός μιας ε, ημερομηνίας 1η Ιανουαρίου 2014 όπως ζητεί η Ζαμβία ή όπως ε, ζητούν άλλοι 1η Ιανουαρίου 2016. Δεν θα είναι λοιπόν δυνατόν να αλλάζει διαρκώς η άποψη και η ημερομηνία και δεν θα μετατίθεται η ημερομηνία εφόσον θα έχει υπάρξει ρύθμιση της τροποποίησης του κανονισμού τελικά. Λοιπόν, εγώ πρότεινα το 2016 ως ημερομηνία. Γιατί πρότεινα το 2016. Εν μέρη επειδή κατανοώ τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι κάποια στιγμή πρέπει να είμαστε συμβατοί και να συνάδουμε με, τα, με τις προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Και θα πρέπει εδώ να δούμε και τα προβλήματα. Δεν δέχομαι ότι υπάρχει μια σημαντική ξεχωριστή περίπτωση έναντι του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για παραβίαση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση των υποχρεώσεών τη και απειλέ ε, να αναλάβουν δράση κάποιε χώρε. Και αν δεν γίνει μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2014, οι χώρε μη ΑΚΕ αναπτυσσόμενε χώρε θα έχουν αρνητική αντίδραση. Δεν λέω ότι θα είναι ικανοποιημένε, ε, δεν υπάρχει τέτοιου είδου ε, ε, προοπτική, αλλά για την ε, τροποποίηση αυτή αναφέρομαι. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι πιθανό θα έπρεπε λοιπόν να, να ευθυγραμμιστούμε με μια ημερομηνία που να είναι συμβατή με τον ΠΟΕ, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Γιατί το 2016, διότι όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με μια μελέτη που χρηματοδοτήσαμε εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο, δεν, είμαστε, δεν προτείνουμε στις χώρες αυτές να απολέσουν την προτιμησιακή αντιπροσωπεία ε, ε, αντιμετώπιση ε, το 2014 Λέει αυτή η μελέτη ότι οι περισσότερες αυτές συμφωνίες ε, σε σχέση με τον Ιούνιο 2012 θα είναι αδύνατο για αυτές τις χώρες να υλοποιήσουν τη διαδικασία επικύρωσης μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2014. Όταν θα φτάσουμε λοιπόν το στο Σεπτέμβριο θα έχουμε ξεπεράσει ήδη αυτό το ορόσημο για να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις αγορές μας τα προϊόντα αυτών των χωρών με προτιμησιακό καθεστώς. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι το 2014 είναι μια θετική ημερομηνία. Επίσης να είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για κάποιο αφηρημένο γενικό λόγο ζήτημα, έχει χειροπιαστέ σημαντικέ επιπτώσει στι χώρε για τι οποίε κάνουμε λόγο. Η Κένια θα είναι ο μεγαλύτερο χαμένο αν υιοθετήσουμε το 2014 ω ημερομηνία θα χάσουν τις δασμολογικές προτιμήσεις ε, για τα αγαθά τους. Ε, ιδιαίτερα για τα φρέσκα, για τα νοπά ε, άνθη, τα λουλούδια που εξάγουν. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, διότι ταυτόχρονα όταν θα έχουμε μηδενικούς δασμούς σε άλλα αγαθά και ξαφνικά θα έχουμε δασμούς που θα πρέπει να καταβάλλονται για τα λουλούδια, θα υπάρξει αντιστάθμιση αντίστροφη σε σχέση με την Κολομβία για παράδειγμα. Θα αντικαταστήσει μία περίπτωση την άλλη. Και όταν έχουμε τα θέματα της Ναμίμπια και της ε, Μποσουάνα, που θα είναι άλλη μεγάλη χαμένη πιθανότητα το πρόβλημα πολύ λιγότερο συνδέεται με την μη προθυμία τους ε, να ευθυγραμμιστούν, αλλά λόγω του ότι αποτελούν μέρος της Τελωνιακής Ένωσης της Μεσημβρινής Αφρικής και πρέπει μέσα στο πλαίσιο της ΣΑΝΤΕΚ αυτής της ε, περιφερειακής οργάνωσης να υπάρξει μια συμφωνία και ρύθμιση. Και ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιείται σε αυτό το πλαίσιο είναι η περιφερειακή ολοκλήρωση. Υπάρχει εδώ το ε, ενδεχόμενο σε σχέση με την Μποτσουάνα ε, να υπάρξει η ευθυγράμμιση αλλά χωρίς να παραβιάσουν την ε, περιφερειακή αλληλεγγύη. Και βλέπουμε ότι για την Αμήμπια 59 εκατομμύρια ευρώ στοιχίζει αυτό σε απώλειες όσον αφορά δασμούς ε, για ε, ηχθιοπροϊόντα και ε, προϊόντα βοηού κρέατος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και άμεσα συνδεόμενο με αυτό το θέμα η Ναμίμπια θα χάσει το 2014 τα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και αυτό θα είναι σημαντικό πλήγμα πάλι εις βάρος της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη. θα έπρεπε να μην δράσουμε και να μην θεωρηθεί ότι δρούμε άδικα και εις βάρος της περιφερικής ανάπτυξης υιοθετώντα την ημερομηνία του 2014. Η Επιτροπή Περιφερικής Ανάπτυξης πρότεινε να μην υπάρξει κάποια τέτοια καταληκτική προθεσμία. Η δική μου πρόταση είναι να έχουμε το 2016 ως καταληκτική προθεσμία. Αν δεν το υιοθετήσουμε αυτό για το επιχείρημά μου, η ομάδα μου δεν θα είναι με κανένα τρόπο υπέρ της 1 Ιανουαρίου 2014. Θα απορρίψουμε τον κανονισμό και δεν μπορώ υπό οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις ε, να επανέλθω στην πρόταση αυτή, να επανεξεταστεί ως ε, ημερομηνία η 1η Ιανουαρίου 2014. Ευχαριστούμε τον εισηγητή μας, ο οποίος ε, έχει ριζοσπαστική θέση για κάθε θέμα. Σκιώδης εισηγητές, ο Κρίστοφερ πρώτα. Κρίστοφερ Φέλνιερ. Ο κύριος Φέλνερ πρώτα. Σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με την προσπάθεια να διαφοροποιήσω κάποια πράγματα. Αναγνωρίστηκε ότι πρέπει να υπάρξει ε, μια καταληκτική προθεσμία σε αυτό το καθεστώς. Από το 2007 η ιδέα ήταν μια προσωρινή λύση για να καλυφθεί ένα κενό που είχε δημιουργηθεί. Το 2007 έως το 2014 είναι αρκετά χρόνια και στις συζητήσεις για το αν χρησιμοποιήθηκε καλά αυτό το χρονικό διάστημα και αν όλοι έδρασαν επικοδομητικά ή όχι. Εμείς πρέπει να βρούμε μια καταληκτική ημερομηνία. Εκεί που δεν συμφωνούμε είναι σε σχέση με την αναφορά για το 2007 και δεν είναι κάτι τυχαίο αυτό. Υπάρχει λόγος και που πρόσφατα ε, ήταν για το 2014. Μετά από την συνεργασία με τα θέματα GSP 1η Ιανουαρίου 2007 είχε αναφερθεί και αν δούμε χώρες ε, όπως το Εκουαδόρ που είχαμε πάμπολες συζητήσεις για τις δικές τους ανάγκες ε, να μπορούν ε, ως χώρα να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα με αυτόν τον τρόπο και μετά να λέγεται ότι αυθαίρετα για κάποιες χώρες, ιστορικές χώρες θα έπρεπε παρότι θα χάσουν την προτιμησιακή αυτή αντιμετώπιση να καταλήξουμε στο 2014, πρέπει να δούμε είναι αυτό δίκαιο ή όχι. Για την Μποτσουάνα για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε την πολιτική μας ε, για το εμπόριο με βάση αυτές τις αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω όμως τις απόψεις ε, των ε, ε, συμβαλωμένων. Αλλά για να ξέρουμε μόνο για ποιο πράγμα κάνουμε λόγο υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις. Τώρα θα πούν κάποιοι πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό ενώ το Εκουαδό δεν θα βρίσκεται σε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχει μια, λοιπόν, μια συγκεκριμένη λογική λοιπόν για το πλαίσιο του 2014. Δεν συμφωνώ με το επιχείρημα που άκουσα από κάποιους φίλους μας της ε, της ομάδας των χωρών ΑΚΕ ότι αυτός ο κατάλογος είναι μια προσπάθεια να τους πιέσουμε και να τους εκβιάσουμε να, να υπογράψουν. Διότι αν υπήρχε ένα ζήτημα σε σχέση με τον ΠΟΕ αυτό δεν θα ε, μπορούσε να γίνει με κανένα τρόπο. Και ρυθμίζοντας έτσι το θέμα με μια καταληκτική ημερομηνία και εμείς θα γνωρίζουμε και εκείνοι τι πρέπει να γίνει. Και αυτό ήταν το χαρακτηριστικό αυτής της συζήτησης. Αν είχαμε μόνο θέματα πρόσβασης ε, στην αγορά θα είχαμε ένα πλούστερο πλαίσιο. Εμείς όμως είχαμε λόγους να μην επιλέξουμε αυτή την ε, προσέγγιση. Η προσέγγιση στην αγορά δεν θα επιτύχει την, δεν θα δώσει την λύση στα θέματα της πολιτικής για την ανάπτυξη. Θα πρέπει να δούμε και τα θέματα των εξαγωγών και του ανοίγματο των αγορών. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε μια διαφορετική θέση να μπορούσαμε να ε, προωθήσουμε τις επενδύσεις. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη όθηση, προώθηση και μεγάλο συμφέρον να υπάρξει ε, μια ταχύτερη ρύθμιση. Ο λόγος για τον οποίο τα κάνουμε όλα αυτά είναι να υπάρξει ανάπτυξη, περιφερειακή ανάπτυξη σε αυτές τις χώρες για την πολιτική ανάπτυξη. Πιστεύω λοιπόν ότι να έχουμε μια συνεκτική πολιτική και να αντιμετωπίζουμε τους εταίρους μας των τρίτων χωρών με δίκαιο τρόπο, νομίζω η πρόταση του 2014 είναι καλή, είναι θετική και για τα δικά μας συμφέροντα και τα δικά, δικά τους συμφέροντα δημιουργεί νομική, ε, νομική βεβαιότητα και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αρθούν τα εμπόδια. Το 2014 εξυπηρετεί λοιπόν και να μην αναμείνουμε κάποια υστερότερη ημερομηνία 2015-2016 τι θα μπορούσε μέχρι τότε και σε ποιο ποσοστό να γίνει και να επιτευχθεί καλύτερα. Γι' αυτό από πλευρά τη ομάδα μα είμαστε υπέρ του 2014 ω ημερομηνία. Και άτυπα έχουμε συζητήσει και έχουμε κάνει την προσπάθεια να βρούμε συμβιβασμού. Καμιά φορά είναι εύκολο να καταλήγει κανεί σε συμβιβασμού. Υπάρχουν κάποια θεμέλια στα οποία μπορεί να χτίσει κανεί μια τέτοια προσπάθεια. Το πρόβλημα εδώ είναι ξεχωριστό και βλέπουμε ότι είναι θέμα ημερομηνία. Ίσως ε, είναι θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί για το πώ θα ψηφιστεί και θα εγκριθεί. Η δική μας πρόταση θα ήταν για την ημερομηνία 2014. Αν δεν περάσει αυτό, τότε θα ψηφίσουμε υπέρ κάποια άλλη χρονική προσέγγισης που θα είναι πολύ κοντά όμω το 2014 και δεν θα απέχει πολλά χρόνια από αυτήν. Νομίζω η καλύτερη πολιτική προσέγγιση είναι αυτή, είναι ο στόχος μας. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε το θέμα. Υποθέτω ότι σήμερα μπαίνουμε περισσότερο στις λεπτομέρειες και γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή για το περιεχόμενο που μας περιέγραψε πάλι. Ποιες είναι οι προκλήσεις δηλαδή Θέλω να είμαι ειλικρινής και σαφής από την αρχή. Εγώ θα προτείνω να απορρίψουμε την πρόταση και υποθέτω ότι δεν εκπλήσεται και ο Φιέλνα για τη στάση μου αυτή και θα σας πω γιατί. Δεν θέλω να συγκρίνω μήλα με αχλάδια. Αλλά θα θυμόσαστε ότι η διάσκεψη του G20 το 2008 με την οικονομική κρίση είπε τα δύο επόμενα χρόνια χρειαζόμαστε ρύθμιση για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση έτσι ώστε να έχουμε μια πιο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Χτες άκουσα τα συμπεράσματα της διάσκεψης κορυφής πάλι των G20 2012, ε. οπότε σχεδόν πέντε χρόνια μετά. Ακόμα όμως δεν υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση. Αν μη τι άλλο όμως υπάρχει συνειδητοποίηση χωρών οι οποίες θα έπρεπε υπεύθυνα να δράσουν για την οικονομική τους ε, ανάπτυξη και δεν μιλάω μόνο για εδώ, μιλάω για ολόκληρο τον κόσμο. Συνεπώς δεν πρόκειται μόνο για εμπορικές σχέσεις. Φυσικά και υπάρχουν εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις αναπτυγμένες χώρες και τις χώρες ΑΚΕ και τις άλλες που μιλάμε. Αλλά εξαρτώνται οι σχέσεις αυτές από την εξέβρεση λύσεων. Οπότε αν σαν αναπτυγμένη χώρα δεν είσαι σε θέση να βρεις μια κοινή ρύθμιση, μια κοινή προσέγγιση για να αντιμετωπίσεις αυτές τις παγκόσμιες προκλήσεις, προφανώς οι διαπραγματεύσεις που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες οικονομικές εξελίξεις των συγκεκριμένων χωρών, στις οποίες αναφερόμαστε, τότε λοιπόν και αυτές θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να συζητήσουν μεταξύ τους και να δουν τι διαπραγματεύσεις θα κάνουν μαζί μας. Οπότε πρόκειται για την ίδια την πραγματικότητα που ισχύει στις χώρες αυτές. Γι' αυτό και καταλαβαίνω πολύ καλά την προσέγγιση του Μάρτιν. Αλλά καταλήγω σε διαφορετικό συμπέρασμα. Ήμουνα με την Επιτροπή μας και εγώ και στην Κένε και στη και τα ακούσαμε τα διάφορα επιχειρήματα. Πήραμε μια ιδέα της πραγματικότητας ε, των χωρών αυτών και πρέπει να συμμεριστούμε τις ανησυχίες μας και με τις ανησυχίες των χωρών αυτών για τις διαπραγματεύσεις. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αν μιλάμε για νέα εμπορική στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και τα συμφέροντα και τι ανησυχίε και των δύο πλευρών. Και των Ευρωπαίων δηλαδή, αλλά και τη άλλη πλευρά, των Αφρικανικών ιδιαίτερα χωρών. Να που μιλάμε και για την Ανατολική Αφρική συγκεκριμένα. Γι' αυτό και πρέπει να δείξουμε ελαστικότητα στις διαπραγματεύσεις. Να σεβαστούμε τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης της κάθε χώρας ΑΚΕ ο κύριος στόχος είναι η προσαρμογή στους κανόνες του ΠΟΕ. Γι' αυτό και δεν πρέπει να πιέσουμε τις χώρες ΑΚΕ να αναλάβουν δεσμεύσεις οι οποίες πηγαίνουν πέρα από το πλαίσιο των συμφωνιών ε, του ΠΟΕ. Μια τέτοια προθεσμία, εφόσον τη βάλουμε τώρα για το 2014, σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει μέσα στο 2012 να ολοκληρωθούν. Λίγοι μήνες μένουν δηλαδή. Άρα πρέπει να επιταχυνθεί και η οικονομική πολιτική στις διάφορες χώρες. Υπάρχουν όμως και αναδυόμενες οικονομίες, οι οποίες μακροπρόθεσμα μπορεί να έχουν μεγάλες προοπτικές και για μας. Τέλος, ο καθορισμός προθεσμίας ε, αντιτίθεται στην αρχή της συνοχής και παραβιάζει το άρθρο 208 της συνθήκης της Λισαβόνας και θα ήταν σε βάρος των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εν λόγω χώρες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εξακολουθεί να ισχύει ο κανονισμός 15-28. Αυτή είναι η θέση μου τώρα και αυτή θα είναι και η θέση μου όταν καταλήξουμε με αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Κέλλερ τώρα. Ευχαριστώ. Αναφερθήκατε στην πολιτική για την ανάπτυξη και ο προλαλή είπε ότι όντω έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αλλά παραβιάζεται το άρθρο 238 της συνθήκης οπότε η συνοχή της πολιτικής πρέπει να είναι στο συμφέρον όλων των πλευρών και να πηγαίνει υπέρ των στόχων ανάπτυξης μεταξύ άλλων της απάλληψης της ένδυας. Αυτό πρέπει να υπάρχει παντού και είναι ένα επιπλέον θετικό σημείο. Αν βεβαίω οι γενικευμένε προτιμήσει είχαν προχωρήσει τώρα όμω, είμαστε σε άλλο επίπεδο. Η Επιτροπή που γνωμοδότησε για την πρόσβαση στην αγορά, η Επιτροπή ΔΕΒΕ, η Αναπτυξιακή, γνωμοδότησε λοιπόν συστήνοντας την Ίντα να μην υπερψηφίσει αυτήν την περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά. Τα επιχειρήματά τους είναι πρώτον ότι η τροποποίηση ε, περιορίζει τις δυνατότητες ολοκλήρωσης στην περιοχή. Και περιορίζει άρα και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσβαση στην αγορά και ο σχετικός κανονισμός θα στρεβλώσει τις εμπορικές ροές. Φυσικά και αντιλαμβάνομαι τα επιχειρήματα ορισμένων ε, αφρικανικών χωρών και άλλων χωρών και που νιώθουν ότι τους ε, βάζουμε έναν εκβιασμό. Απ' την άλλη, αν δεν έχετε πιστεί από τα επιχειρήματα υπέρ της ανάπτυξης, ακούστε κάποια προβλήματα που υπογραμμίστηκαν από το Think Tank η e CDPM που είναι ένα think tank εδώ στις Βρυξέλλες που γνωρίζει πολύ καλά η Επιτροπή, συχνά ε, ενημερώνεται. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα πράσινο οργανισμό. Και λέει ότι υπάρχουν προβλήματα με την πρόταση της Επιτροπής και πιο συγκεκριμένα ε, εντοπίζουν δύο ζητήματα. Πρώτον, λένε το άρθρο 230β λέει ότι μπορεί να αποσύρει το δικαίωμα στην αγορά μόνο όταν δεν έχει υπάρξει επικύρωση σε ένα λογικό χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση, άπαξ και έχουν αναλυφθεί βήματα. Συνεπώς, πρέπει να μην έχει γίνει η επικύρωση μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Ωραία, δεν έχει γίνει. Στην πρότασή της λέει ότι δεν έχουν αναλυφθεί ε, βήματα, τα οποία όμως δεν φτάνουν για να γίνει και επικύρωση, χρειάζεται κάτι παραπάνω. Δεν υπάρχει δηλαδή για μένα νομική βάση εδώ. Δεύτερο πρόβλημα, υπάρχουν και άλλα, λόγω θα περιοριστώ σε αυτά τα δύο, λέτε η πρόταση της Επιτροπής έχει και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα. Ο καθονισμός 1528 είναι μια μονομερής διάταξη εφαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι εξαρτάται από την ε, σύμβαση της Βιέννης που μιλάει για την εφαρμογή τέτοιων συμβάσεων. Οι προϋποθέσεις δεν ικανοποιούνται. Μια λοιπόν που πρόκειται για μια εφαρμογή μονομερή εμπίπτει στα πλαίσια της ε, σύμβασης της Βιέννης όπου αναφέρονται διάφορες προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να γίνεται ο περιορισμό αυτός που θέλουμε και που δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον έτσι λέει το Think Tank. Η μελέτη αυτή δεν είναι καινούρια. Είναι το Οκτωβρίου του 2011. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τη γνωρίζει και θα ξέρει τι προβλήματα αναφέρει. Οπότε έχουν κάποια απάντηση σε αυτό. Πάντως δεν πρόκειται απλώ για πολιτικά επιχειρήματα θέλω να πω για την πρόσβαση στην αγορά. Υπάρχουν νομικά ζητήματα που μπαίνουν στην περίπτωση που γίνει αυτή η τροποποίηση. Πρόεδρος, ε, η συνάδελφος Πέρντεν, ο πρόεδρος ε, σήμερα το πρωί μας πρότεινε ε, να καθορίσουμε από μόνοι μας πώς θα συνεχίσουμε με τις προεδρίες. Συνεπώς τώρα που θα πάρει το λόγο η συνάδελφος θα δώσω στον συνάδελφο Λάγκια την προεδρία. Θα φύγω εγώ και ο επόμενος εκ περιτροπής προεδρία, δηλαδή σήμερα. Και ίσως θα έπρεπε να το κάνουμε πάντα αυτό. Ίσως να μπει και καμιά γυναίκα στο Προεδρείο καμιά φορά, κύριε Πρόεδρε, τι λέτε. Ο τίτλος είναι πολύ ενδιαφέρον. Μιλάει για συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Αλλά εγώ δεν βλέπω και πολύ εταιρική σχέση. κάποια στιγμή στις διαπραγματεύσεις τη λέμε, λέμε ορίστε έχετε δύο μήνες. Το μήνυμα ακούστηκε δυνατά και ξεκάθαρα. Και επιπτώσεις έχει. Γιατί πάρα πολλοί νιώθουν ε, τώρα άβολα, νιώθουν να απειλούνται και υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια εξαιτίας ε, της ρύθμισης αυτής που προτείνουμε. Ίσως θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερη διπλωματία και πιο μετρημένα και πιο πολύ βάση της εταιρικής σχέσης να προχωρήσουμε. Πολλά ακούστηκαν για την προσέγγιση η οποία ήταν πάντα να στηρίζουμε την περιφερειακή συνεργασία. Και κυρίως στην περίπτωση της Ανατολικής Αφρικής όπου μπορεί να καταλήξουμε να βγει η Κένια από τις συμφωνίες, αυτό θα αποσταθεροποιούσε την περιοχή πολύ σοβαρά. ως ζώνη ελεύθερου εμπορίου θα δείτε ότι τελικά θα πηγαίνουν προϊόντα στην Ουγκάντα και από εκεί θα φεύγουν. Θα υπάρξει αποσταθεροποίηση αν πιέσουμε τόσο πολύ και βιαστούμε χωρίς να είναι όλοι έτοιμοι για αυτή την εταιρική σχέση. Όντως, περνάει ο καιρός. Σωστά. Εγώ ακούω από τους συναδέλφους της συνεδριάσης ΑΚΕ ότι η Επιτροπή αλλάζει τους στόχους. Δεν ξέρω αν ισχύει. Πάντως δεν ε, τους αρέσει βέβαια. Και πρέπει να το πούμε. Το ότι δεν έχουν υπογράψει τίποτα δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει και τίποτα. Έπειτα, για μας δεν είναι εύκολο από εδώ να καταλάβουμε πως τα Υπουργεία μιλούν με εξωτερικούς εταίρους, αλλά όχι με την υπόλοιπη κυβέρνηση, ίσως με τα άλλα υπουργεία. Είναι πολύ εσωστρεφή. Και δεν τα λένε με την υπόλοιπη κυβέρνηση απαραίτητα. Και αυτό βέβαια δημιούργησε πρόβλημα όταν έφτασε η προθεσμία. Συνεπώς, το μήνυμα έχει ακουστεί. Το βάλαμε το ζήτημα και το ακούσανε. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι κάνουν και εκείνοι και όπως λέει και ο Ντέβι, το 2014 προκειμένου να προχωρήσει ολόκληρη η νομοθεσία δεν φτάνει ο χρόνος. Οπότε εφόσον υπάρχει μια ημερομηνία, θα είναι ικανοποιημένο. Νομίζω λοιπόν ότι καλό είναι να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια περικοπή, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να μπορεί να εφαρμοστεί. Το 2016 με ικανοποιεί, θα υπάρχει χρόνος ακόμα. Ε, ε και ακόμα και όταν ε, τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα, στις διαπραγματεύσεις χάνεται χρόνος. Νομίζω ότι η πρόταση είναι λογική, ε, πρέπει να είναι και επικοδομητική ταυτόχρονος ε, και επομένως να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο τις διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα δεν έχουν ζητήσει άλλη τον λόγο. Γι' αυτό θα δώσω τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και η συνάδελφος, η κυρία Γκαλίνα, Head of Unit, θα πάει τον λόγο. Thank you. Good morning, Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Πολύ σύντομα. Θα ξεκινήσω αποσαφηνίζοντας κάποιες παρατηρήσεις, κάποια θέματα. Η συζήτηση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Καταδεικνύει ακόμα ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι απόλυτα σαφή σε σχέση με την πρότασή μας. Ξεκινώντας η εξαίρεση waiver του ΠΟΕ Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για παράδειγμα υπό την προτιμησιακή αντιμετώπιση του Βάμβακα το 2001 ε, εγκρίθηκε εκπνέει το 2007 δεν έχουμε τώρα καθεστώς τέτοιας εξαίρεσης. Βρισκόμαστε στο 2012 και συζητούμε ακόμα αν θα έχουμε το 2014 ή υστερότερα μια χρονική στιγμή για την καταληκτική αυτή ημερομηνία. Τα επιχειρήματα αυτού του κανονισμού ήταν απλά, ήταν μια γέφυρα που δημιουργούσαμε. Αναγνωρίζετε ότι ήταν πολύ δύσκολο το 2007 να επικυρωθούν όλα αυτά από τις ε, χώρες και αποφασίσαμε ότι μονομερός θα προχωρούσαμε με το πιο γενναιόδωρο καθεστώς ε, που θα προσφέραμε από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, χωρίς δασμολογικές επιβαρύνσεις για τα προϊόντα βάμβακα, χωρίς να επιβαρύνονται από πλευράς μας αυτές οι χώρες. Ένα έτος, δύο έτη. Αυτό ήταν αρχικά εκείνο το οποίο σκεπτόμαστε ότι θα υπαρκούσε για την επικύρωση. Το πολύ τρία χρόνια. Αλλά το 2014 θα ήταν ε, πάνω από έξι χρόνια Κάπως εκπλήσωμε λοιπόν πρέπει να πω ότι εξετάζουμε και να έχουμε ιστερότερη ημερομηνία μετά το 2014. Δεν θα αναφερθώ στην νομική αβεβαιότητα και ανασφάλεια που θα ε, συνεπαγόταν κάτι τέτοιο όσον αφορά τις επιπτώσεις για την πολιτική, για την ανάπτυξη, που δεν θα υπήρχαν ε, επενδύσεις ε, και δεν θα γινόντουσαν επενδύσεις επειδή δεν θα υπήρχε νομική βεβαιότητα και ασφάλεια για αυτές τις χώρες. Έχουν ε, επιλογή εναλλακτική αυτές οι χώρες. Μπορούν να επικυρώσουν τις συμφωνίες, τις συμφωνίες είτε αυτές που μονογραφήθηκαν είτε υπογράφηκαν στο παρελθόν. Μπορούν σχετικά γοργά να προχωρήσουν και θα υπάρχει αρκετός χρόνος από σήμερα μέχρι το 2014 για να το πράξουν αυτό. Θα έλεγα ότι κάποιες χώρες προτιμούν να επιλέξουν κάποιες άλλες συμφωνίες ε, περιφερειακής εμβέλειας, ε, ευρύτερης, ε, μεγαλύτερου εύρους και για λόγους ευελιξίας είπαμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντάξει ωραία μπορούμε να αναμείνουμε να υπογραφούν και να επικυρωθούν αυτές οι συμφωνίες και μπορώ να σας πω ότι οι διαπραγματεύσεις βαίνουν αρκετά καλά. Εκπλήσωμαι από την πολύ αρνητική εντύπωση που έχετε όλοι αποκομίσει για κάποια αίσθηση για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να, να χαρακτηριστούν οι διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή. Ως προς αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι παρότι αυτό το οποίο αποκαλείται ε, μεμονωμένο θέμα, παρότι κάποια από αυτά τα μεμονωμένα θέματα συζητώνται απλά, απλά και μόνο, μόνο μετά από αίτημα αυτών των ε, συμβαλωμένων εταίρων. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ευρύτερα πλαίσια και αυτό είναι ένα παράδειγμα ευελιξίας και ελαστικότητας. Μπορώ να σας δώσω πολλά άλλα παραδείγματα μέσα από ένα μεγάλο κατάλογο αυτής της ευελιξίας. Να θυμόσαστε ότι δεν, δεν δημιουργούμε δεν δημιουργούμε εμπόδια και προσκόμματα με κανένα τρόπο στις διαπραγματεύσεις μας με αυτές τις χώρες. Αν θέλουν να διαπραγματευτούν κάποιες χώρες, πολύ καλά να το κάνουν. Μπορούν να το κάνουν, διαφορετικά δεν υπάρχουν προβλήματα. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι οι εταίροι μας είναι αρκετά ικανοποιημένοι. Θα έλεγα, μπορούν λοιπόν να επικυρώσουν την προηγούμενη συμφωνία, μπορούν να επιλέξουν να ε, επικυρώσουν την ε, επόμενη ή μπορούν και να θέλουν εντάξει, να αντιμετωπίζονται ως οποιαδήποτε άλλη χώρα, αναπτυσσόμενη χώρα. Και ως προς αυτά η πρόταση λοιπόν δεν θα έχει επιπτώσει στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες οι εννέα λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες θα βρισκόντουσαν υπό το καθεστώς τα πάντα εκτός από όπλα, everything but arms. Κάνουμε λόγο για δύο χώρες λοιπόν, Μποτσουάνα και Ναμίμπια που θα μπορούσαν να εκπέσουν, να βρεθούν εκτός αυτού του πλαισίου. Όλες οι άλλες ε, έξι αναπτυσσόμενες χώρες αν απεμπολίσουν αυτό και δεν είναι αυτό το οποίο βλέπω να γίνεται γιατί θέλουν να συνεχίσουν είτε με τη νέα συμφωνία είτε με την επικύρωση της παλαιότερης. Και έτσι θα υπάρχει η δασμολογική προτιμησιακή αντιμετώπιση των προϊόντων τους. Αυτό πρέπει να δούμε. Γυρνώντας η σελίδα σε σχέση με τα ωφέλη που θα υπάρχουν θέλουμε να υπάρχει σαφήνεια σε σχέση με τέρους μας από τις χώρες ΑΚΕ. Κανένας δεν μπορεί, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την Ευρώπη ότι δεν ήταν γενναιόδορη. Κανείς, μα κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Να το θυμόμαστε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τους δώσαμε χρόνο, τους δώσαμε επαρκές χρονικό διάστημα και βοηθάμε αυτές τις χώρες να ξεπεράσουν ακόμα και τα πιο μικρά εναπομείναντα εμπόδια. Έτσι λοιπόν με αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτή την προσέγγιση πρέπει να αντιμετωπιστούν οι διαπραγματεύσεις μας και η προοπτική μας. Θα ήθελα επίσης να πω ότι νομικά δεν κάνουμε λόγο για κάποια εφαρμογή. Τα θέματα αυτά θα μπορούσαμε διμερώς να τα συζητήσουμε. Αλλά θέλω να σας διασφαλίσω όλους σας ότι η, προτάση, η πρόταση από νομικής πλευράς είναι απόλυτα στεγανή θα έλεγα. Είναι απόλυτα καθαρή, κοσέρ θα ήθελα να μας υποστηρίξετε για μια πολύ ισόρροπη, ισορροπημένη προσέγγιση από πλευρά μας. Είναι ισόρροπη και ισορροπημένη αυτή η προσέγγιση. Προσπαθώ να προσπαθούμε να εντάξουμε όλους, προσ, ε, μεταθέτοντας την τελική ημερομηνία, καταληκτική ημερομηνία στο 2014. Είναι πραγματικά μια γενναιόδορη ε, χειρονομία από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περίμενε 10 χρόνια και παραπάνω για να ρυθμιστεί αυτό το θέμα. Και κατανοώ ότι υπάρχουν κάποια θέματα, αλλά κανείς δεν μπορεί, κανείς να κατηγορήσει ότι δεν είμαστε γενναιόδοροι. Ευχαριστώ. Yeah, Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλερ, μια υπερώτηση παρακαλώ. Μόλις είπατε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την νομιμότητα του θέματος. Μπορείτε να μας τα εξηγήσετε λίγο γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία ανέφερα και σημαντικό και ενδιαφέρον θα ήταν να πούμε αν τα προβλήματα, να δούμε αν τα προβλήματα που ανέφερα είναι ε, ορθά υφιστάμενα ή όχι και θα ψηφίσουμε πότε, το απόγευμα όχι αύριο ε, και πριν ψηφίσουμε χρειαζόμαστε σαφήνεια. Κύριε Γελίνα. Καλό είναι να είμαστε σαφείς λοιπόν. Θα είμαι... Θα... Λοιπόν, ε, πρόνοια πρόνοιες της ε, Συμφωνίας Γουιάννα προβλέπει ότι και από την άλλη πλευρά θα υπάρχει κάποια... Ε, ε, ε κάποια αμοιβαιότητα και βλέπω ότι τώρα μόλις ξεκινάει κάτι τέτοιο και το λέω μα Λοιπόν, με τον κανονισμό για την πρόσβαση στην αγορά, αυτό που κάναμε ήταν μόνο μερός, και το τονίζω, μόνο με μονομερός ε, να προχωρήσουμε σε ε, εφαρμογή της συμφωνίας η οποία δεν αναγνωρίστηκε από την άλλη πλευρά. Η, στη συνθήκη της, Βιέννα, της Βιέννης ε, ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει αμοιβαιότητα και από την άλλη πλευρά και ξέρετε ότι και βάσει του άρθρου 25 ε, ε, ε, ανεφέρει κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Βιέννης που μου είναι ιδιαίτερο γνωστή δεν γίνεται κάτι ξαφνικά. Εμείς όμως το κάναμε για λόγους καλής θελήσεως και καλή την πίστη. Ε, λοιπόν, μονομερός αποφασίσαμε να διευρύνουμε ε, την ε, διάταξη αυτή χωρίς μάλιστα και σύμφωνη γνώμη του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, πράγμα όχι πολύ σορθό. Μετά από το 2017 δεν υπάρχει καμία κάλυψη πλέον και επομένως αυτή η μονομερής πράξη τελικά δεν είναι αμφισβητήσιμη από νομικής απόψεως αλλά ταυτοχρόνως νομίζω ότι αυτή ήταν και η πολιτική βούληση και δεν καταργούμε λοιπόν το ε, προτιμησιακό καθεστώς. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Και ο εισηγητής ο ίδιος θα λάβει τώρα τον λόγο για να ολοκληρώσει παρακαλώ. Thank you to... Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους και την Κομισιόν. Δεν θα απαντήσω βέβαια σε όλα τα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν, σε ορισμένα μεταξύ αυτών. Βεβαίως μπορεί να πει η Κομισιόν ότι από το 2007 δεν έχουμε τη σύμφωνη γνώμη ε, του Παγκοσμίου ε, Οργανισμού Εμπορίου. Δεν μίλησα βέβαια με, όλους, τι όλες τις χώρες ε, του ΠΟΕ, μίλησα όμως με εκπροσώπους των κάποιων από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ξέρω τις ανησυχίες τους όταν προκύπτουν ζητήματα, καμία χώρα μέχρι τώρα δεν μου έχει κοινοποιήσει την πρόθεσή της να αναλάβει οποιαδήποτε ε, δράση. Επιπροσθέτως και κάτι που ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι. Εάν ε, ε, πάρουμε απόφαση για το 14, το 17 ή το 19, τότε θα, θα καθησυχαστούν τα πνεύματα. Εγώ συμφωνώ με την ανάλυση του ε, Helmet, αλλά ε, νομίζω ότι η πρώτη επιλογή μπορεί να είναι διαφορετική. Δεύτερο σημείο και δεν θα μπω σε όλες τις λεπτομέρειες Νομίζω ότι μπορούμε να γνωρίσουμε το σχόλιο της Επιτροπής σχετικά με το ε, κατά πόσον πρέπει ή μπορούμε να πιέσουμε τους ε, ε, συνομιλητές μας να δεχτούν τη συνθήκη της Σιγκαπούρης και να πω ας πούμε ότι όταν πήγαμε στην Κένια είχαμε ε, briefing της Κομισιόν που μας έλεγε ακριβώ αυτά και μετά μιλήσαμε με τον ε, επικεφαλής ε, των διαπραγματεύσεων από πλευράς της Κένιας και εν πάση περιπτώσει μας είπε ότι όλα τα συζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά όταν ξαναπήγαμε στην Κομισιόν ε, μας είπε ναι εντάξει τα βάζουμε στο τραπέζι για αυτά τα ζητήματα για να τα, να τα συζητήσουμε αλλά δεν πιέζουμε και πάρα πολύ έτσι ώστε να προωθηθούν πρέπει να ξέρουμε ε, τι είμαστε προετοιμασμένοι να διαπραγματευτούμε, πόσο, ε, πόσο θα προωθήσουμε την διαπραγμάτευση επιορισμένων ε, θεμάτων κλπ. και οδηγούμε λοιπόν σε αυτό που είπε ο Κρίστοφερ. Δεν λέω ότι ορισμένα από αυτά τα θέματα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περισσότερο και ότι δεν θα μπορούσαν να, να πέσουν στο τραπέζι. Υπάρχει όμως σημαντική διαφορά ε, ανάμεσα στη διαπραγμάτευση καλών συμφωνιών για αυτά τα θέματα ή ε, απλά να διαπραγματευτεί κανείς την πρόσβαση στην αγορά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα όταν ε, ανοίξουν αυτά τα κεφάλαια τότε χρειάζεται πραγματογνωμοσύνη και επιμονή έτσι ώστε να ολοκληρωθούν. Σε σχέση με αυτά που ακούσαμε από την Κομισιόν, θέλω να πω το εξής οι επιλογές των χωρών ΑΚΕ, ε, ναι βεβαίως η επικύρωση είναι ε, μία ε, επιλογή. Δεν το κάνω επίτηδες, αλλά ξέρω την Κένια καλύτερα ενδεχομένως. Εάν η Κένια, ας πούμε, προσυπογράψει, επικυρώσει και κάποιες γειτονικέ χώρες της Ανατολικής Αφρικής δεν υπογράψουν, τότε θα βρεθεί αποκομμένη από την ε, περιφερειακή αγορά. Οι χώρες της Ανατολικής ε, ε, Αφρικής είναι χώρες οι οποίες εμπίπτουν στο Everything But Arms και επομένως θα πρέπει να δούμε αν θα υπογράψουν όλοι. Μιλήσαμε εκτός, με από την Κένια και με άλλους εκπροσώπους άλλων χωρών και αυτές οι άλλες χώρες έχουν και λίγο διαφορετική γνώμη και ε, και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς ε, πιέζεται η Κένια να πάρει ε, μία θέση έτσι ώστε ένα μέρος του εμπορίου τελικά των εμπορικών συναλλαγών τελικά ε, να οδηγηθούν προς τις ε, γειτονικές χώρες. Ε, κάποια στιγμή όλα αυτά θα πρέπει να τελειώσουν, να σταματήσουν και πιστεύω ότι θα πρέπει να βάλουμε στόχους επιτεύξιμους. Γι' αυτό μιλάω για το 16 και όχι για το 14. Ευχαριστώ. Είναι σαφής η σύσταση του εισηγητή. Αύριο θα ψηφίσουμε γι' αυτό και θα λάβουμε έτσι απόφαση. Νομίζω είναι δίκαιο για την πλειοψηφία να στείλουμε έτσι ένα σαφές μήνυμα στους εταίρους μας. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε έτσι το σημείο 8 στην ημερήσια διάταξη. Περνάμε στο 9. Δραστηριότητες εποπτικής ομάδας, monitoring group, ομάδων εποπτικών. Το βρίσκω σωστό και σημαντικό επανειλημμένα και πάντα να έχουμε αναφορά του τι γίνεται ώστε αυτές οι εποπτικές ομάδες να μην παρεκκλίνουν πολύ σημαντικά από τις δραστηριότητες της κοινοβουλευτική μας επιτροπής και αποκτήσουν ξεχωριστή δική τους αυτοσύστατη ζωή και γι' αυτό έχουν συνεδριάσει εντωμεταξύ και μόνο μία υποπτική ομάδα συνεδρίασε, εμείς συνεδριάσαμε, μόνο μία ομάδα υποπτική συνεδρίασε για την Κεντρική Αμερική η υποπτική ομάδα. Δίνω τον λόγο στον μόνιμο εισηγητή μας για να μας πει τα σχετικά από αυτή τη συνάντηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για την τελευταία συνεδρίαση της εποπτικής ομάδας που προέδρευε ο ίδιος γιατί η δική μου πτήση ακυρώθηκε και δεν μπορούσα την προηγούμενη Δευτέρα να είμαι στις Βρυξέλλες. Θα ήθελα να σας επεξηγήσω σύντομα την κατάσταση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Κεντρικής Αμερικής. Αποφασίστηκε τελικά η Επιτροπή Εμπορίου να έχει δύο εμπόρια, δύο εκθέσεις που θα ε, έχει αφενός για το άρθρο 50 και το δεύτερο για την συνενετική συνενετική διαδικασία για τη συμφωνία. Η Κορεπέρ θα δώσει αύριο την σύμφωνη γνώμη, όπως προβλέπετε, και στις 25 του μήνα δεν είναι το Συμβούλιο που θα εγκρίνει. Έτσι και στις 28-29 Ιουνίου αυτού του μήνα πάλι επίσης προβλέπεται η υπογραφή της ε, συμφωνίας στην Τεγκουσιγκάλπα, πρωτεύουσα τη Ορδούρα. Έχουμε ένα σχέδιο λοιπόν που πρέπει να συντονιστεί και να ε, ε, συγκεκριμενοποιηθεί με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Να υποβληθούν και τα δύο κείμενα είναι η ιδέα από πλευρά του άρθρου και τη συμφωνία και στι 12 Ιουλίου στην ε, δική μα Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα παρουσιαστούν και θα έχουμε κατάθεση τροπολογιών με καταληκτική προθεσμία όπω θα αποφασιστεί και στην Επιτροπή ΙΝΤΑ τον Σεπτέμβριο θα επανεξεταστεί και τον Οκτώβριο θα δοθεί συνέχεια για την ψήφιση και έγκριση από κοινού τα δύο έγγραφα της ε, ίντα και για την ε, συνένεση για τη συμφωνία και για την ρήτρα διασφάλισης ε, δικλείδα ε, δικλίδα ασφαλείας. Σε μία από τις Ολομέλειες του Σεπτεμβρίου θα ε, ψηφιστεί η προσέγγιση. Η νομική μας υπηρεσία αναγνώρισε, ε, εντόπισε κάποια οριζόντια προβλήματα νομικού χαρακτήρα που αφορούσαν και τις δύο συμφωνίες συμπεριλαμβανομένης και αυτής της συμφωνίας ΕΕ Κεντρικής Αμερικής. Φαίνεται ότι ευτυχώς υπάρχει η βούληση πολιτική βούληση και θεσμική βούληση, κυρίως από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να εξευρεθεί μια λύση που θα είναι αποδεκτή για μας που σίγουρα θα συμπεριληφθεί στις παραγράφους για την δικλίδα ασφαλείας, για τη ρήτρα ασφαλείας. Προβλέπετε να επιληθεί χωρίς ε, κάποια προβλήματα. Έτσι λοιπόν, αν έχετε κάποια ερώτηση, είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος που να ζητά τον λόγο. Όμως κύριε Σιγητά, ίσως θα μπορούσατε και πάλι να μας πείτε ποιος είναι ο συσχετισμός ε, ε, του θέματος αυτού όσον αφορά τη ρήτρα διασφάλισης, τη δικλίδα ασφαλείας, διότι ακριβώς αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή τη συμφωνία και την ρήτρα ασφάλειας, δικλίδα ασφαλείας και θα ήταν η βάση αυτή για μια ε, προσέγγιση. Ευχαριστώ. Πράγματι, όσον αφορά τις ρήτρε, προβλέπετε να ψηφίσουμε στις 12 Ιουλίου τις τροπολογίες εδώ στην Επιτροπή αυτή. Στη συνέχεια θα έχουμε τριμερείς διαλόγους και θα ψηφίσουμε τη ρήτρα τον Οκτώβριο. Η βασική ιδέα είναι η ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή μας ίντα να γίνει παράλληλα με την ψηφοφορία στην Ολομέλεια για να καθησυχαστούμε ότι οτιδήποτε κρεμότητα κλείνει. Ja, yeah, good. Μάλιστα, πολύ καλά. Λοιπόν, Ολοκληρώνουμε εδώ αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Επόμενο σημείο είναι η συνάντηση των συντονιστών μας και κλεισμένων των θυρών. Παρακαλώ όλοι όσοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετάσχουν να εγκαταλείψουν την αίθουσα.